Colleagues, if I can ask you all... Παρακαλώ, καθίστε. Ούτω ώστε να συνεχίσουμε την απογευματινή μα συνεδρίαση, Σήμερα να ξεκινήσουμε την απογευματινή συνεδρίαση και να συνεχίσουμε την πρωινή. Λοιπόν, πρώτος συντονιστής που έχουμε είναι ο κ. Βαλέντε Ντε θα μας μιλήσει για τους αυτοκινητόδρομους της θάλασσας. Πρόγραμμα 21. Λοιπόν, ας καθίσουμε. Μία μόνο συνεδρίαση σε αυτή την αίθουσα, όλες οι άλλες εκτός παρακαλώ. Okay. So. Λοιπόν, κύριε Βαλέντα Ντολιβέρα, είχατε το λόγο για κάνα δεκάλεπτο να μας εξηγήσετε περί τίνος πρόκειται όσο αφορά το πρόγραμμα 21 και μετά θα υποβληθούν ερωτήσεις και θα ακουστούν σχόλια από τα μέλη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς συγχαρητήρια για την θέση που αναλάβατε. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Θα μιλήσω πορτογαλικά τώρα. Αν επιτρέπετε βέβαια. Κανένα πρόβλημα λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, τα τελευταία δύο χρόνια είχα συναντηθεί με διάφορους ανθρώπους για να ετοιμάσουμε αυτή την έκθεση η οποία συζητείται. Αυτή είναι η δεύτερη. Η πρώτη υπευλήθη πέρσι από Φιλανδία μέχρι Ελλάδα. Ξετάσαμε τα λιμάνια και τα δρομολόγια. Πρόκειται για σειρά λιμανιών και διαμετακόμισης, αλλά και λιπάνια που κάνουν τις ε, transshipment και interland, τις δύο αυτές ε, διαδικασίες. Ε, λοιπόν, Αναφερόμαστε λοιπόν στο θέμα των σκαφών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τα διάφορα συστήματα που χρησιμοποιούν όπως συστήματα VTS και άλλα και το φορτίο των σκαφών και τον εξοπλισμό του και το πλήρωμα. Αυτό το είχα καλύψει στην πρώτη ε, έκθεση. Έχουμε πρώτα απ' όλα τα πλοία μεταφοράς φορτίου, τα container ships. Συζητούσαμε το θέμα της βελτίωσης των μεταφορών. Να υπάρχουν μικρότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και πώς, τι ισχύ χρησιμοποιούν οι κινητήρες, οι μηχανές των σκαφών και πώς μπορούν να διασυνδεθούν τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα. Όσον αφορά τις μεταφορές, μιλάμε και για τη σύνθεση των πληρωμάτων όσον αφορά τα σκάφη. Τρεις χώρες στην Ευρώπη δεν έχουν προβλήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης των πληρωμάτων. Η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Νορβηγία, που δεν είναι βεβαίως μέλος της Ένωσης. Όλοι οι άλλοι έχουν πρόβλημα κατάρτισης και εκπαίδευσης των πληρωμάτων και νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε τον ενδεχόμενο ως προγράμματος τύπου έρασμους για την εκπαίδευση των πληρωμάτων. Λοιπόν, αποτελεσματικότητα των λιμανιών είναι η δεύτερη ομάδα προβλημάτων από διοικητική σκοπιά. Σε πρώτερη έκθεσή μου επικεντρώθηκα στην ενία θηρίδα. και μπορούν να γίνουν πάρα πολλές βελτιώσεις διοικητικές. Πολλών ειδών υπηρεσίες μπορούν να καλυφθούν και να συμπεριληφθούν και η αποτελεσματικότητα, η υποδοτικότητα ενός λιμένος εξαρτάται από αυτό. Η επόμενη ομάδα προβλημάτων είναι πραγματικά φυσικά προβλήματα. Κάποια λιμάνια πρέπει να ε, αυξήσουν το βάθος που έχουν. Μετά είναι το θέμα του εξοπλισμού. Θέσεις δεν υπάρχουν αρκετές για τα πλοία. Για να βελτιωθούν λοιπόν τα λιμάνια αυτά πρέπει να τα λύσουμε. Κυρίως τα λιμάνια που είναι σε πόλεις και περιβάλλονται από την υπόλοιπη πόλη, κυρίως όταν η πόλη είναι πολύ παλιά πόλη και η επέκταση της πόλης περιορίζεται λόγω του λιμανιού. Άρα μπορούν να γίνουν πολλά όσον αφορά και τον εξοπλισμό των ε, λιμάνιων. Στην είσοδο του λιμανιού πολύ συχνά πρέπει να πληρούνται διάφορες προϋποθέσεις για να μπορεί το πλοίο να μπει και πρέπει να είναι σαφής η όρη που θα καλύπτουν όλα τα λιμάνια. Αυτές οι είσοδοι είναι πάρα πολλές σημαντικές. για να μπορέσουμε να καθορίσουμε διάφορους δείκτες που θα χρησιμοποιούμε για, τον, ε, για τους υπολογισμούς μας και την ενιαία θηρίδα. Θέλουμε δείκτες, παραδείγματος χάρη, για την αποδοτικότητα των λιμανιών. Όλα αυτά τα στοιχεία που παρέθεσε είναι σημαντικά. Μετά θέλουμε να δούμε τι γίνεται με την ενδοχώρα. Τους σιδηροδρόμους θα θέλαμε να χρησιμοποιούμε γενικά για πρόθεση των εμπορευμάτων στην ενδοχώρα. Εγώ υποστηρίζω για τη μείωση των καθυστερήσεων και για να είμαστε αποτελεσματικοί όσον αφορά τη χρήση των σιδηροδρόμων να βελτιώσουμε την κατάσταση. Να μην συμβαίνει αυτό που είδα πολύ συχνά στην Πολωνία και στη Ρουμανία. Τι συμβαίνει δηλαδή, τι πρέπει να αποφύγουμε. Υπάρχουν χρειάζονται αυτοκινητόδρομοι, ε, χρειάζεται κάποιο μήκος και, ε, αυτοκινητόδρομο για να συνδέσει το λιμάνι με την ενδοχώρα. Οι διασυνδέσεις με την ενδοχώρα χρειάζονται κάποια μέρημνα από πλευράς Ένωσης. κυρίως από πλευράς επιμελητίας και οργάνωση γενικά. Πριν από δύο εβδομάδες πήγα στο Bremerhaven και εκεί υπάρχουν διασυνδέσεις με την ενδοχώρα και πολύ αποτελεσματικές διασυνδέσεις και μπόρεσα να δω τι λύσεις χρησιμοποιούν εκεί και θα ήθελα αυτό να γίνει συνήθεια σε όλα τα λιμάνια, σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν όλη η αλυσίδα της επιμελητίας να αναλυθεί. Να εξετάσουμε όλη την αλυσίδα των μεταφορών, πώς λειτουργεί. Πριν προχωρήσω σε συγκεκριμένες συστάσεις που έχω συμπεριλάβει στην έκθεσή μου, θα ήθελα να σας πω και το εξής. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει ένα συντονισμό των πολιτικών σε διάφορους τομείς. Θα μπορούσα να παραθέσω πάμπολα παραδείγματα. Σχέση μεταξύ μεταφορών και περιφερειακής πολιτικής, παραδείγματος χάρη, μεταφορών και έρευνας. Μεταφορών και τελωνίων. Ο συντονισμός αυτών των τομέων είναι πάντα πολύ δύσκολος. Αλλά ίσως θα έπρεπε να γίνει ένα συντονισμό σε ζευγάρια, αν δεν είναι δυνατό να καλύψουμε τα πάντα και να καλύψουμε τρεις-τέσσερις πολιτικές ταυτόχρονα. Γι' αυτό υποβάλλω σχετικά κάποιες συστάσεις, θα τις διατρέξω εντάχει. Έχω 12 σημεία. Αναφέρομαι στην ολοκληρωμένο χαρακτήρα των λιμανιών, βελτίωση των διασυνδέσεων με την ενδοχώρα και το τονίζω, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πολιτική μας. Ανοιχνευσιμότητα των σκαφών πάρα πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου και πισμός αυτών η ανάπτυξη ευραίων, ευραίου φάσματος μελετών διότι χωρίς μελέτες ε, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά γι' αυτό χρειάζονται μελέτες το υπογραμμίζω αυτό διότι πάντα αμφισβητούμε την αξία των διαφόρων μελετών που διαθέτουμε. Αν θέλουμε να συγκρίνουμε κάποια πράγματα, να συγκρίνουμε τα λιμάνια, παραδείγματο χάρη, πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μα και τις κατάλληλε μελέτες από κάπου να αντλήσουμε στοιχεία για τη σύγκριση. Η βελτίωση τώρα των σχέσεων μεταξύ των λιμανιών και των συναφών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το λιμάνι. Η εκπαίδευση των πληρωμάτων. Από διοικητική πλευρά η ενιαία θηρίδα, η έρευνα και ανάπτυξη, πολύ σημαντικό στοιχείο και οι διασυνδέσεις μεταξύ διαφόρων πόρων, διαφόρων χρηματοδοτήσεων. Αυτό που ανακάλυψα και πιστεύω ότι ήταν καλό είναι ότι υπάρχουν ε, διάφορες μορφές χρηματοδοτήσεως. Έχουμε το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Περιφερειακής Αναπτύξεως, το πρόγραμμα Μάρκο Πόλο, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Οι εταίροι μας δεν ξέρουν ποιο φορέα να χρησιμοποιήσουν, σε ποιον να αποτανθούν για να ζητήσουν χρηματοδότηση. Γι' αυτό είναι σημαντικό και το προτείνω αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει ένα συμβουλευτικό σύστημα, ούτως ώστε ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση στις κατάλληλες πληροφορίες. χρειάζεται για και απλούστευση της γραφειοκρατίας, επικαιροποίηση των στοιχείων, απλούστευση της γραφειοκρατίας κυρίως στις Βρυξέλλες και κάτι καινούριο το οποίο θα ήθελα να θίξω. Νέες σχέσεις με γειτονικές χώρες, νέες διασυνδέσεις με γειτονικές χώρες και με συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας με τα οποία έχει επαφή, έχει σχέση η Ευρώπη. Τι εννοώ με αυτό που λέω. Διασυνδέσεις με την Άπο Ανατολή. Μερικές, μερικά δρομολόγια περνάνε το Σουέζ, άλλα δρομολόγια περνούν από τον Παναμά. Άρα δεν μπορούμε να διαφορούμε για αυτά που σημαίνει στον Παναμά ή στο Σουέζ. Και είναι πολύ σημαντικό για την μελλοντική μας ευμάρεια αυτά να τα προσέξουμε. Εν τέλει, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη στατηγική σημασία των θαλασσίων μεταφορών. Όπως προανέφερα, ταξίδεψα πολύ, επισκέφθηκα διάφορα λιμάνια και είδα ότι τα διάφορα μέρη έχουν διαφορετικά προβλήματα. Άλλα προβλήματα έχει η Αδριατική, έχει πολλές δυνατότητες η Αδριατική που δεν χρησιμοποιούνται, η Βυρική Χερσόνησος έχει προβλήματα, ο Εύξηνος Πόντος έχει προβλήματα αλλά προσφέρει και πολλές προοπτικές και ίσως λύσεις για διασυνδέσεις με άλλα μέρη του κόσμου και αυτά πρέπει να τα εξετάσουμε. Και βέβαια και οι διασυνδέσεις Ανατολής με Δύση, διαμέσου της Μεσογείου. Αυτές οι διασυνδέσεις έχουν τεράστια σημασία για την Ευρώπη. Η Άπο Ανατολή βέβαια είναι στην οθόνη του ραντάρ μας. Είναι πολύ δυναμική περιοχή, αλλά έχουμε και τη Λατινική Αμερική, όπως η Βραζιλία. Έχουμε χώρες της Αφρικής που θα μπορούσαν να μας ενδιαφέρουν και μπορούμε να εξετάσουμε το θέμα. Λοιπόν, αυτά έχω να πω πάρα πολύ σύντομα για την έκθεση μου, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ερωτήσεις και ομιλητές. Από το ΕΛΚ ο κύριος Ήταλα. Σωστά το πρόφερα. Σωστά το προφέρατε. Ευχαριστώ. Συμφωνώ. Ε, άποψή μου η εισαγωγή ήταν εξαιρετική. Το σχέδιο αυτό των θαλασσίων ε, αυτοκινητοδρόμων είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έρχομαι από τη Φιλανδία. Είμαστε στην άκρη της Βαλτικής και αυτό το, αυτός ο διάδρομος για μας είναι πολύ σημαντικός. Το πρόβλημα είναι ότι προχωρά αργά και είμαι βέβαιος ότι θα υλοποιηθεί μεν, πότε όμως δεν είναι ένα ανοιχτό ερώτημα πρέπει να προχωρήσει ταχύτερα η χρηματοδότηση του έργου για να έχουμε απτά αποτελέσματα. Επίσης, να ζητήσω από το συντονιστή, να θέσω μια ερώτηση στον συντονιστή. Μιλάμε για την ενιαία θηρίδα. Έχετε υπόψη στο φιλανδικό σύστημα. Το σύστημα της ενιαίας θηρίδας στη Φιλανδία έχει δουλέψει σωστά και έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του. Επίσης, ασφάλεια στη θάλασσα στη Βαλτική υπάρχουν πάρα πολλά σκάφη, ρωσικά πολλά από αυτά, που τηρούν διαφορετικές διατάξεις από εμά και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για να επιβάλλουμε στους Ρώσους να τηρήσουν κάποιους κοινούς, κάποιες κοινέ διατάξεις. Περιβάλλον τώρα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός μίλησε για την ανάγκη μείωσης των εκπομπών θείου πριν το 2015, ούτω ώστε να μειωθεί το ποσοστό εκπομπών από το 0,5 στο 0,1. Δεν ξέρουμε τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στο κλίμα, αλλά αποτελεί μια τεράστια θυσία για την οικονομική ε, δραστηριότητα τα σκάφη με τον στόχο αυτό δεν θα μπορέσουν να, να λειτουργήσουν. Στη Φιλανδία μόνο μια τέτοια αλλαγή των καυσίμων θα οδηγήσει σε αύξηση των δαπανών της ναυπηλίας κατά ένα δις μόνο για την ε, Φιλανδία. Για την, ε, υπάρχουν οι χώρες ε, οι εταιρείε θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό αυτό, η Σουηδία, η Stena Lines, ενώ από την άλλη Έχουμε τους Ρώσους που συνεχίζουν να ρηπαίνουν χωρίς πρόβλημα και θα κερδίσουν επιπλέον. Πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί μία λύση που είναι, γιατί το πρόβλημα είναι σοβαρό για όλα τα κράτη. Η μείωση από 0,5 σε 0,1 είναι καταστροφικό για την Φιλανδία. Ο κύριος Στέρξ. Ευχαριστώ πρόεδρε. πάντα απορούσα τι ακριβώς είναι αυτά τα αυτό το τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων γιατί στους σιδηροδρόμους, στον αυτοκινητόδρομο, ακόμη και στο κανάλι που θα κατασκευάσουμε καταλαβαίνουμε λίγο πολύ περί τίνος πρόκειται. Εδώ πέρα ομολογώ ότι πάντοτε μου φαίνονται ασαφή τα στοιχεία Και βλέπω δυστυχώς επίσης ότι κανένας, κανένα μεγάλο εγχείρημα δεν επέτυχε. Μήπως θα πρέπει να υποβάλλετε και πάλι την ε, ερώτησή σας. Ναι, αφού λοιπόν δεν με καταλαβαίνετε πολύ καλά, να σας πω. Λέτε ότι έχουν επιτύχει τα μεγάλα σχέδια κτλ. Βεβαίως, για το συντονιστή. Η κριτική είναι κάπως σκληρή. Καταλαβαίνω ότι αυτά που μας λέτε για τα λιμάνια ότι είναι πολύ σημαντικά, ότι η λειτουργία τους είναι καλή, ότι υπάρχουν καλές υποδομές, ναι, ωραία. Αλλά όταν υπάρχει μεταφόρτωση εμπορεύματος από το ένα πλοίο ε, και ε, μάλλον για το, όσον αφορά τη μεταφόρτωση εμπορεύματος ε, από ένα πλοίο σε άλλο μέσο, πολύ καλά. Πλην όμως πρέπει να πω ότι σε ένα σεμινάριο που ήμουν εγώ για τις θαλάσσιες οδούς, ή καλύτερα για από το αυτοκινητοδρόμους, ετέθη ζήτημα εάν θα ξεκινούσαν και προγράμματα υποδομών και αν θα έπρεπε να υπάρχουν τερματικοί σταθμοί πολύ λειτουργικοί στους οποίους θα έπρεπε να ε, δοθεί κάποια υποστήριξη, τουλάχιστον για την εκκίνηση της ανάπτυξής τους. Και από την άλλη υπάρχουν κάποιες ε, γραμμές που έχουν απτυχθεί μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας, αλλά η χώρα στηρίζεται μόνο στην ε, υποστήριξη από τις κυβερνήσεις. Μετά υπάρχει και το άλλο το θέμα των eco-bonus από την Ιταλία, όπου ένας ε, μεταφορέας θα εξασφάλιζε ένα bonus, ένα πριμ, εφόσον ε, επέλεγε όχι τη συνοδική μεταφορά, αλλά την διαφαλές μεταφορά εμπορευμάτων την διαφαλέ μεταφορα εμπορευματων απο το ένα στο άλλο λιμάνι της Ιταλίας. Μπορεί να δουλέψει ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε κάποιες λύσεις ε, αποτελεσματικές πιστεύετε. Για μένα δεν είναι καθόλου ξεκάθαρη αυτή η εικόνα. Τι σημαίνει αυτοκινητόδρομος της θάλασσας και τι μπορεί να προσφέρει επιπλέον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα να ζητήσω να μου πει ο συντονιστής πώς έχουν τα πράγματα για τον διάδρομο 21 στην Αδριατική και τι προβλέπετε για τις χώρες ε, της Βαλκανικής δεδομένων του τι έγινε και τι συμβαίνει. Ε, επίσης υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια αύξησης της ποταμοπλοείας στον Πάδο. Προβλέπετε να υπάρξει σύνδεση του πάδου με το σύστημα, με το διάδρομο 21. Ευχαριστώ, Τέμπορα. Από το ΕΛΚ, τη Τσιέρα, τη Σέιρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να σημειώσω ότι ήταν μεγάλο προνόμιο και τιμή για μένα το ότι είχα την ευκαιρία να δω εδώ τον ε, Πορτογάλο προγνώμονα και να ακούσω τις ε, πληροφορίες που είχε να μας δώσει με βάση την εμπειρία του. Ε, σημειώνω ότι δεν χρειάζεται να υπογραμμίσουμε τη μεγάλη σημασία των δρομών της θαλάσσης για κράτη, περιφερειακά, ε, όπως η Πορτογαλία και ιδιαίτερα η Μαδέρα, η δική μου ε, ιδιαίτερη πατρίδα. Χρειάζεται λοιπόν οι θαλάσσιες μεταφορές για να αναπτυχθούν, να αποτελέσουν μια ε, εναλλακτική, να μετατραπούν σε μια εναλλακτική λύση ανταγωνιστική. Το λιμάνι του Σίντσι παραδείγματι στην Πορτογαλία θα μπορούσε με εμβάθυνση να ε, αξιοποιηθεί γιατί είναι αρκετά ρηχό τώρα και να αποτελέσει ένα καλό λιμένα ε, και πολυλειτουργικό ακόμη. Εδώ η διασύνδεση με άλλους τρόπους μεταφοράς έχει τεράστια σημασία ασφαλώς και χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ορατότητα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ως προς τους αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας. χρειάζεται μια διαφορετική διαμόρφωση των ε, ε, αυτοκινητοδρόμων της θάλασσας και δυνατότητα μετάβασης, διαλειτουργική δηλαδή αξιοποίηση σε άλλα μέσα μεταφορών. Αυτές είναι οι προτάσεις μου, αυτές είναι οι ιδέες που θα ήθελα και να σας ρωτήσω συγκεκριμένα ποιο ε, στοιχείο μπορεί να παίξει τον καταλητικό ρόλο ε, για την επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Βρεξελών αφενός και τοπικών περιφερειακών αρχών. Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το σχέδιο αυτό ώστε να ρονταριστεί και να πάρει ταχύτητα ε, πλεύσης. Η κυρία να έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ από πλευράς μου να ευχαριστήσω τον ε, ομιλητή μας για τις εξηγήσεις μας έδωσε για τις προτάσεις του, την έκθεσή του. Και να πω ιδιαίτερος ότι πρέπει να εξετάσουμε την πρόσβαση στις ε, θάλασσες, ιδιαίτερα για τη Βαλτική επί παραδείγματι. Βλέπουμε ότι οι εφοπλιστές έχουν αναλάβει δράση πληθωρική θα έλεγα. Δηλαδή δεν μας λείπουν ε, οι εφοπλιστές, δεν λείπουν τα καράβια. Δεν υπάρχει αρκετός χώρος, δεν υπάρχουν αρκετά, ε, αρκετές χερσαίες οδοί που να πηγαίνουν προς τα λιμάνια για να αξιοποιήσουμε τα λιμάνια μας. Τι είδους λοιπόν υποδομές πρέπει να αναπτύξουμε κατά την άποψή σας για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους εφοπλιστές μας και πώς πρέπει να αναπτυχθεί η υποδομή μας έτσι ώστε να διατηρηθεί αδιάκοπη μία ε, αλυσίδα επιμελητιακή. Επίσης, ε, στον προϋπολογισμό για τους αυτοκινητοδρόμους της θάλασσας, στο Μάρκο Πόλο, ε, έχετε κάποιες συγκεκριμένες προτιμήσεις, α το πω έτσι, οι επιθυμίες, κάτι που θα θέλατε οπωσδήποτε να αναφέρετε, που θα μπορούσαμε εμείς να συμβάλλουμε ως αρχή αρμόδια και για τον προπολογισμό, έτσι ώστε να προβλεφθεί κάτι συγκεκριμένο με την ευκαιρία των νέων δημοσιονομικών προπτικών από το 2013 δηλαδή και έπειτα. Επίσης ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε και νωρίτερα, στη σχέση μας ε, με την Ρωσία εδώ έχουμε να κάνουμε και με την, ε, με την ε, Βαλτική ασφαλώς, ε, αλλά και με, την, με τη Μαύρη Θάλασσα, με τον Εύξηνο Πόντο. και συμφωνίες μεταφορών. Εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε καλύτερη επικοινωνία, επαφή και λειτουργία αυτών των συμφωνιών ε, και των εμπορικών φυσικά συναλλαγών με τη Ρωσία, έτσι ώστε ε, χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις να μεταφέρονται τα προϊόντα, αλλά να μεταφέρονται κατά προτίμηση και από θαλάσσιες, έτσι ώστε να έχουμε ώστε δυνατόν λιγότερη ρήπανση. Εδώ νομίζω ότι το, το Gateway to the Sea νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία και ασφαλώς θα πρέπει να το εξετάσουμε και αυτό ως λύση Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Βάισνερ είναι ο τελευταίος Κυρία. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον κύριο Ολιβέηρα. Πολύ σύντομα, για να συμφωνήσω με τα όσα ακούστηκαν νωρίτερα, όπως είπε και ο Φινλανδός συνάδελφος, υπάρχει ήδη το πρόβλημα της επιβάρυνσης με θείο με μόλιβο όσον αφορά τα καύσιμα που χρησιμοποιούν αυτά τα πλοία ε, και ίσως χωρίς βέβαια να είναι ιδεώδης λύση αυτή να μπορέσουμε να μειώσουμε τις, ε, την περιοκτικότητα σε μόλιβδο αν και θα πρέπει να φροντίσουμε τα μέτρα που θα εισαχθούν να είναι μετρημένα έτσι ώστε να μην ε, χρειαστεί να μεταφερθούν εναλλακτικά δηλαδή των θαλασσινών μεταφορών, τα προϊόντα αυτά μέσω των σιδηροδρόμων ή των αυτοκινητοδρόμων, πράγμα το οποίο θα επιβάρει ακόμη περισσότερο το περιβάλλον μας. Επίσης, σε σχέση με λιμάνια τα οποία ε, ε, βαθύνονται και μπορούν να λάβουν και εμπορεύματα ή να συνδεθούν διαλειτουργικά ε, με άλλες περιοχές, ε, πώς μπορούμε να προωθήσουμε ένα σχέδιο με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά ένα τέτοιο σχέδιο. Ευχαριστώ. Και αν μου επιτρέπετε κύριε Ολιβέηρα. για τις ε, γραμμές των θαλάσσιων μεταφορών και την, ε, τον κανονισμό του της Εθνούς Οργάνωσης Ναυτιλίας το 2015 γιατί θεωρούν ότι είναι 0,1% το ποσοστό που μπορούμε να περιμένουμε βάσει των προβλέψεων αυτής της οργάνωσης ε, για τις ε, μικρών αποστάσεων θαλάσσιες μεταφορές. Ίσως θα έπρεπε αυτό να το δούμε κάπως ε, πιο προσεκτικά, κυρίως το γεγονός ότι παραδόξως πώς έχει αποκλειστεί η Μεσόγειος από τους υπολογισμούς αυτούς. Θέλετε παρακαλώ να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους ε, βουλευτές για τις ερωτήσεις τους. Ας ξεκινήσω με τη Φινλανδία πρώτα, την οποία έχω επισκεφθεί. Έχω επισκεφθεί το Κότκα και το Χάμινα, δύο λιμένες, όχι το Ελσίνκι δηλαδή, ε, που έχω επισκεφθεί εγώ και ασφαλώς γνωρίζω πόσο δύσκολα η γεωγραφικά είναι η περιοχή και ποιες είναι οι ευαισθησίες σχετικές με το πετρέλαιο κακής ποιότητας από τη Ρωσία ή με πολύ θείο που προέρχεται από περιοχές ή μάλλον που περνάει από περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες και έτσι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της συνεργασίας, μάλλον τη διάρθρωση σε σχέση με τη Ρωσία γιατί ο μεγαλύτερος χώρος συγκέντρωσης ε, της κατανάλωσης στη Ρωσία, μεταξύ δηλαδή Αγίας Πετρούπολης και Μόσχας, είναι περίπου 70 με 80 εκατομμύρια ε, πολίτες που έχουν υψηλό υψηλή αγοραστική δύναμη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε λύσεις ε, οι οποίες έχουν να κάνουν είτε με την επιλογή της Βαλτικής, με το σχετικό κίνδυνο, είτε μέσω είτε ε, από το βόρειο παγωμένο ε, ωκεανό με, παγοθραυστικά, είτε φυσικά η καλύτερη λύση θα ήταν ένα οργανωμένο, ολοκληρωμένο, πληρέστερο σύστημα. Για την ε, πύλη τώρα, το gate που εκπροσωπούν το Gothenburg και το Άρχους, ασφαλώς θα ήταν μια καλή λύση για να αποφευχθεί η διέλευση πλοίων που δεν χρειάζεται εξάπαντος να περάσουν από εκεί ή πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνες ή που αποτελούν τα ίδια ε, κίνδυνο στις μεταφορές. Συμφωνώ λοιπόν ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες για τα νέα σκάφη ιδιαίτερω πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση και συμφωνώ και με εσά κυρία μου για τις ανησυχίε που εκφράσετε για το θείο, για την περιεκτικότητα σε θείο και χρειάζομαστε καλύτερες, ε, καλύτερους κινητήρες, καλύτερα σκάφη και όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Συμφωνώ επίσης ως προς τις τοποθετήσεις ε, τις σχετικές με την πειθαρχία που απαιτείται για τα παλαιότερα σκάφη και δεν θεωρώ ότι είναι καλή λύση ή μάλλον καλή εφεύρεση οι σημαίες ευκαιρίας. Οι σημαίες ευκαιρίες, ευκαιρίες ή τα σκάφη που προέρχονται, που έχουν σημαία κράτους, όχι τόσο υπεύθυνου ως προς την ναυσιπλοεία, όχι τόσο σοβαρού, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, να διωχθούν θα έλεγα, με ε, διεθνή συνεργασία. Για τους αυτοκινητόδρομους της θάλασσας, κύριε Στέρκ, ε, η δυσκολία είναι ότι δεν είναι ορατή ταυτόχρονα, δεν είναι ορατές ταυτόχρονα οι τρεις συνιστώσεις στις οποίες αναφέρεστε. Δηλαδή δεν βλέπουμε σκάφος, λιμένα και hinterland ταυτόχρονα, ενδοχώρα δηλαδή ταυτόχρονα. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να προετοιμαστούμε έτσι ώστε να ε, προετοιμάσουμε την διασύνδεση μεταξύ αυτών των παραγόντων πρέπει, ε, νομίζω, μπορούμε τουλάχιστον θα πρέπει να αποφύγουμε τον, ε, την στρέβλωση του ανταγωνισμού η οποία είναι τόσο σημαντική που την ε, συμπεριέλαβα στην ε, δεύτερη μου έκθεση και θα πρέπει νομίζω να πούμε ότι εάν κάνουμε κάτι στο Αλμάνια ή στο Χίντερλαντ ε, σε σχέση με το Χίντερλαντ θα πρέπει αυτό να γίνει βέβαια σε συνεργασία και με την ε, προοπτική για την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτή είναι η άποψή μου. Κάνατε μια αναφορά Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε σε μερικά χρόνια να έχουμε πείσει και τις εταιρείε. Το ECO-Bonus είναι καλή ιδέα. Η Ιταλική κυβέρνηση καταβάλει μόνο το εξωτερικό κόστος στη μεταφορά. Δηλαδή λέει στο μεταφορέα περάσεις οδικός, σου κοστίζει τόσο. Εμείς σου διαθέτουμε αυτό το ποσό για να χρησιμοποιήσεις το πλοίο. Σου καλύπτουμε δηλαδή με μέρος του κόστους. Αυτό βέβαια και ασφαλώ και εγώ θα ήθελα να δω να επιλύεται το πρόβλημα αυτό είναι ότι καλύπτεται η διαφορά του κόστου στην Ιταλία μένα αλλά όχι μέχρι και την Ισπανία ή την Ιταλία. Και πρέπει να δούμε να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων, τέτοιων δράσεων. Επίσης, θα ήθελα να σημειώσω ότι ήμουν ε, στην ε, Τριέστη, έχω επισκεφθεί τη Τριέστη και άλλες ε, πόλεις, το Κόπερ, τη Βενετία. Και πρέπει να πω ότι στη Βενετία Φερρυπίν έγινε μια τελετή θα έλεγα συνεργασίας υπόσχεση δόθηκε στην τελετή αυτή για συνεργασία μεταξύ των τεσσάρων λιμένων στην Αδριατική. Ένα πράγμα στο οποίο ε, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε, να δώσουμε έμφαση εδώ είναι ότι Υπάρχουν βεβαίως και υπάρχουν δυνατότητε γεωγραφικέ. Βέβαια, η ιστορική δεσμίσεω, μάλλον η ιστορία μπορεί να δημιουργεί κάποιε δυσκολίε και ανησυχίε. Αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξει εν τέλει αυτή η διάρθρωση και θα διασκεδαστούν όποιες υποψίες δυσπιστία υπάρχει μεταξύ των πόλεων αυτών, των λιμένων αυτών. η Ραβένα, η Βενετία, το Μομφαλκόν, η Τριέστη, το Κόπερ και η Ραγέκα είναι η Ριέκα, Κροατία δηλαδή, είναι οι λιμένες που πρόκειται να συνδεθούν. Η Κροατία ήδη έχει ενταχθεί στο σχέδιο αυτό. για την ε, διασύνδεση της Βενετίας με την Κρεμόνα μέσω του Πάδου ε, νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα γιατί ήδη έχουμε το λιμένα μέσα στην ε, Βενετία ήδη υπάρχει η δυνατότητα δηλαδή, διασύνδεσης μέσω του Πάδου από, πλευράς, από την άκρη της Βενετίας και νομίζω ότι μπορούν οι αρχές να μας βοηθήσουν. Και έτσι έχοντας εσωτερικές πλωτές οδούς μπορούμε να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε σημαντικά την κατάσταση. Και ιδιαίτερα να να ενισχύσουμε το ρόλο του ε, λιμένα, της έννοιας του λιμένα, στη Βόρεια Αδριατική. Το ΣΥΝΣ, πορτογαλικό λιμάνι, κοντά στη νοτιο στη νοτιοδυτική πλευρά, ακτή της ε, Πορτογαλίας. Σαντ Βίνκτ που ήταν γνωστός μεγάλος λιμένας Ευρώπης. Ένα λιμάνι λοιπόν ε, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ξεκινήσαμε με βάθος 70 και τώρα έχουμε 35 μόνο μέτρα βάθος. Και έχουμε και πολύ χώρο για επέκταση. Οι λιμένες δεν προτιμούν να είναι μόνο λιμένες ε, μεταφόρτωσης. Με εξαίρεση στον στην Μεσόγειο. Οι λιμένες προτιμούν εν είναι με, ε, λιμένες μεταφόρτωσης και διασύνδεσης με την ενδοχώρα. Το ΣΥΝΣ είναι ένα λιμάνι που χρησιμοποιείται ως ε, λιμάνι μεταφόρτωσης. Θα ήθελε να γίνει λιμάνι ενδοχώρας και να διασυνδεθεί με την Μαδρίτη, η οποία έχει ξηρό λιμένα και πιστεύουμε ότι αν επιληθούν τα προβλήματα θα έχουμε πολύ καλή ε, διασύνδεση του Σύνους με τη Μαδρίτη. Επίσης μιλήσατε για το ρόλο των περιφερειακών ή τοπικών αρχών, των εθνικών αρχών ω προς την ανάπτυξη της σημασία των λιμένων ε, των θαλάσσιων λιμένων. Εγώ πιστεύω ότι η απάντηση είναι καλές μελέτε, καλές προτάσεις, καλά σχέδια και αν είναι καλές οι προτάσεις ασφαλώ, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καλυφθούν οι προτάσει αυτέ με τα απαραίτητα κονδύλια. Για την κυρία Γένσεν. Συμφωνείτε νομίζω κι εσείς για τη σπουδαιότητα να δώσουμε έμφαση στην υποδομή. Πιστεύω ότι τα πράγματα είναι, πάνε αργά. Το είδατε και το πρωί για μια σειρά έργων σιωδρομικού χαρακτήρα ότι καθυστερούν. Χρειάζεται 10-12 χρόνια και παραπάνω ακόμα. καταλαβαίνετε ότι με δεδομένο το ότι ο αριθμός των εμπλεκόμενων είναι πολύ μεγαλύτερο στις ε, θαλάσσιες διασυνδέσεις θα υπάρξουν περισσότερα προβλήματα. Οι νέες χρηματοοικονομικές προοπτικές θα παίξουν ρόλο. και τα λιμάνια και η ενδοχώρα και οι πλατφόρμες επιμελητίας αν αποκτήσουν πρόγραμμα θα βοηθήσουν στην ταχύτερη υλοποίηση. Αλλά, το είπα και προηγουμένως, εάν προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας και χρησιμοποιήσουμε τους διάφορους πόρους και δώσουμε, προσφέρουμε συμβουλευτική στους χρήστες, επιτρέποντας και το να ξεκινήσουν δικές τους πρωτοβουλίες, πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε γρηγορότερα. Νομίζω ότι κάλυψα το ερώτημα με τη Ρωσία. είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε την παροχή εμπορευμάτων από το βορρά προς νότο. Το θέμα της Μαύρης Θάλασσας, της Κωνσταντζας και των βουλγαρικών λιμένων. Επιπλέον έχουμε και το ζήτημα των δαρδανελίων, ενός πολύ στενού διαδρόμου που πρέπει να παίξει ρόλο στην, απάντηση, στην μορφή απαντήσεων που θα δώσουμε. Κύρια Μέσνερ, έχω πάει στο Χάβεν. Ήταν σαφές ότι το νέο λιμάνι που αναφέρεται στο δυτικό τμήμα της πόλης θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Το λιμάνι του Bremenhaven είναι πολύ καλό παράδειγμα συνεργασία με άλλα λιμάνια. Δεν το ξέρει ο κόσμος, αλλά έχουν πολύ καλή συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα ιταλικά λιμάνια, την Gioia Tauro. Και έχουν μία εμπειρία συνεργασίας 30 ετών με συμφωνία με την Τζόια Τάουρο. Αυτό είναι η μορφή απάντησης που χρειαζόμαστε. Συνεργασία μεταξύ πολύ αποτελεσματικών λιμένων και πολύ καλά ε, και λιμένων που βρίσκονται σε πολύ καλές τοποθεσίες. Αυτό είναι νομίζω κάτι που στο οποίο θα πρέπει να προσβλέπουμε στο μέλλον. Για σας τώρα. το πρόβλημα που αναφέρετε, δεν έχω πάει ακόμα στην IMO ή θα τους επισκεφθώ στο Λονδίνο αλλά το πρόβλημα που αναφέρατε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ήθελα να είμαι πιο θετικό στην απάντησή μου, αλλά προ το παρόν όχι. Πάντω ούτε σε όλε θα του επισκεφθώ. Το, το έχω προβλέψει ήδη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βαλέντιντ Ολιβέηρα για την παρουσίαση και τι απαντήσει που δώσατε. Πώς βλέπουμε στην συνέχιση της συνεργασίας μαζί σας στο μέλλον. Λοιπόν, συνάδελφοι, αλλάζουμε το όνομα και ζητώ από την Κάλα Πέις να έρθει να κάτσει δίπλα μου. Δεν φανταζόμουν ότι θα την έβλεπα ποτέ να καθόμαστε δίπλα-δίπλα, πάντως ε, χαίρομαι που σας βλέπω ξανά. Κάρλα. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι τα έργα 18 και 30 εσωτερικές, θαλάσσιες, ε, εσωτερικές πλωτές οδοί Δούναβης και Σκάλδης Καλωσορίζω την Κάρελα στην Επιτροπή. Όλους τους καλωσορίζαμε, αλλά φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε πως η... το καλώς είναι πολύ πιο ειδικό προς την Κάρελα. Έχεις το λόγο, Κάρλα. Ευχαριστώ, Μπράιαν. Καταρχάς να ευχαριστήσω Θα μπορούσα να είμαι ο συντονιστής του εαυτού μου αυτό το καιρό, γιατί ξέρετε ε, στην Ολλανδία υπήρχε μια σύγκρουση μεταξύ των Ολλανδόφωνων και των, των Ολλανδών και των Φλαμανδών, αλλά το πρόβλημα θα λυθεί φαντάζομαι κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ξεκινώ με το τέλος. Να σας πω ποια είναι τα συμπεράσματα που έχω μετά το τέλος του δεύτερου έτους της θητείας μου συντονίστριας. Και μετά να σας ακούσω να μου πείτε αν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Πρώτον, η εσωτερική ναυσιπλοεία μπορεί να είναι η βάση για να αναπτυχθεί και να προωθηθεί μία περιοχή. Η στρατηγική λοιπόν της λεκάνης του Δούναβη θα βοηθήσει την ανάπτυξη της περιοχής γύρω από το ποτάμι. Αντί λοιπόν να βλέπουμε μόνο τον ποταμό, εμείς κοιτάμε την λεκάνη του Δούναβη. Διότι είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί η λεκάνη με όλα όσα γίνονται το ποτάμι. Διότι αν έχουμε ένα ποτάμι πλωτό αλλά δεν έχουμε πλατφόρμες διασύνδεσης ή σύνδεση με βιομηχανικούς χώρους, αν δεν έχουμε προετοιμάσει τα λιμάνια που σχολίασε ο κύριος Ολιβέηρα, τότε θα έχουμε κάνει πολύ κακή δουλειά. Η λεκάνη λοιπόν του Δούναβη είναι το κομμάτι που κοιτάμε δεν είναι μόνο το ποτάμι αυτό αυτό. Αν δείτε λοιπόν την λεκάνη, θα δείτε ότι περιλαμβάνει μια σειρά διαστάσεων κοινωνικών, πολιτικών, περιβαλλοντικών κλπ. Χρειαζόμαστε λοιπόν διαλειτουργικότητα και μετά τις προτάσεις που κάναμε για την ε, μετατροπή του ποταμού σε πλωτό, πρέπει να κοιτάξουμε και την αγορά. Υπάρχει στόλος, πόσος είναι καλός για να καλύψει τις απαιτήσει των τις περιβαλλοντικές απαιτήσει. Το σωστό χρησιμοποιούν, το σωστό καύσιμο. Είναι καθαρά πλοία, πράσινα σε εισαγωγικά συνδέουμε με το ποτάμι του σωστούς βιομηχανικούς χώρους. Συνεργαζόμαστε πολύ με τις αρχές κοινών δηλώσεων, που είναι μια συμφωνία μεταξύ όλων των Υπουργών Περιβάλλοντος των εμπλεκομένων χωρών. Πολλές είναι αυτές για το Δούναβι. Όλες οι κυβερνήσεις συμφώνησαν για αυτές τις αρχές της κοινή δήλωσης και προσθέσαμε και κάτι, διότι αυτό που βλέπουμε στην περιοχή είναι να παλεύουν οι χώρες αυτές με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που θα θέλαμε να δούμε είναι πολύ νωρίς να υπάρξει μια ομάδα ειδικών που θα πηγαίνουν σε μια χώρα όταν εμφανίζεται ένα νέο σχέδιο και θα λένε στις κυβερνήσεις πώς να αντιμετωπίσουν την περιβαλλοντική νομοθεσία. Και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η ομάδα των Πρασίνων, οι, οι ομάδες ε, που προστατεύουν τον περιβάλλον παλεύουν πολύ για το, την προστασία του και, και δίκιο έχουν. Το ποτάμι δεν είναι ένα κάτι άψυχο, είναι μια ζωντα, ένα ζωντανός οργανισμός για τον κόσμο. Ε, υπάρχει ένα τραγούδι που λέει ένα, ε, σε κάθε άνθρωπο υπάρχει ένα ποτάμι. για μένα είναι ο Σκάλβης. Εγώ, για μένα είναι ο Μέρσεϊ, λέει ο πρόεδρος. Για τον κόσμο που μένει κοντά στο Δούναβη, ο Δούναβης είναι ένα ζωντανό, ένα ζωντανός οργανισμός και πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε ως ζωντανό οργανισμό. Θέλουμε λοιπόν να προσφέρουμε ειδικού που έγκαιρα θα πούν στις κυβερνήσεις αν κάνεις αυτό και αυτό με αυτό το αποτέλεσμα, τότε θα σέβεσαι την νομοθεσία. Πρέπει να λύσουμε τα βασικά προβλήματα, τα bottlenecks, αλλά και να λύσουμε τα προβλήματα αν δεν υπάρχουν σκάφη, αν δεν υπάρχει αγορά, αν δεν υπάρχουν λιμάνια, αν δεν υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας των μεταφορέων, λέω που να καταλάβουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν και τα πλοία, όχι μόνο τα φώτιγα, ε, δεν κάναμε τίποτα. Και νομίζω ότι ο Ναϊάντε μπορεί να μα βοηθήσει λίγο, γιατί και αυτό κοίταζε για την πραγματικότητα. Επίση, μα βοηθά πολύ η τεχνολογική εξέλιξη και στις ε, και στις νέες μορφές και, στις νέες, ε, και στα νέα, στις μαούνες και στην τεχνολογία χρήσης. Η γενική εικόνα πάντως αυτή είναι που θα σας δείξω. Πολύ συγκεκριμένα τώρα. Ο δεύτερο χρόνο προχώρησε γρήγορα. Είχαμε πολλέ αλλαγέ κυβερνητικού χαρακτήρα στην Ανατολική Ευρώπη. Και ξέρετε αυτό έχει και πρακτικές συνέπειες. Δηλαδή όταν είσαι συντονιστής και αλλάζει η κυβέρνηση, πα στην κυβέρνηση, του λε: Γεια σα, είμαι αυτό, θέλω να σα βοηθήσω. Και αν κάθε τρει και λίγο αλλάζουν οι κυβερνήσει, ε, δεν είναι εύκολο αυτό. Πήγαμε πολλέ, κάναμε πολλά ταξίδια στις διάφορες ε, παραδουνάβιες χώρες, Βουλγαρία, Ουγγαρία, ε, Ρουμανία. Τον επόμενο χρόνο θα πάμε και σε χώρες που δεν είναι στην Ένωση, παραδείγματος χάρη τη Σερβία. Ευτυχώς, δεν έχουμε μόνο αυτά τα δύο έργα ε, που είναι, που, όπου υπάρχει ενδιαφέρον για την εσωτερική ναυσιπλοεία δηλαδή το Δούναβι, Ρίνο και τον ε, Σικουάνα Σκάλδη και άλλες χώρες, ε, Ιταλία, Τσεχία ενδιαφέρονται. Το πρόγραμμα Ναϊάδες τώρα είναι πολύ σημαντικό γιατί σχετίζεται με το γενικότερο θέμα της ναυσιπλοείας οι πληροφορίες ε, ασφάλειας στο ποτάμι προσφέρουν βεβαιότητα στους ε, εμπλεκόμενους. Ξέρετε, πολλά ποτάμια περνούν από το κέντρο πόλεων και όταν έχεις ε, μεταφορά αγαθών πρέπει να κοιτάξεις και τι γίνεται στις ακτές. Αργότερα θα μιλήσω για την προσέγγιση, έτσι, την μακροπεριφερειακή προσέγγιση. Το, να ξεκινήσω από το, με το γερμανικό πακέτο από βορρά προς νότο. Το γερμανικό κομμάτι είναι το, η περιοχή μεταξύ Στράουμπεν και Βίσχοβεν στη Βαφαρία. Πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο τμήμα Εμείς εδώ θελήσαμε απλά να εφαρμόσουμε τις κοινέ αρχές. Η... Έχει γίνει μια μελέτη από την Βαβαρία και την κεντρική κυβέρνηση, η οποία παρακολουθείται από μια ομάδα παρακολούθησης, στην οποία μετέχουν όλοι τα εμπορικά μελητήρια. Παλιά 30 χρόνια δεν μίλαγε ο ένας τον άλλον. Τώρα μετέχουν όλοι στο ίδιο... Είναι στην ίδια τράπεζα συζητήσεων, σε αυτή ίδια, στην ίδια ομάδα. Τι θέλω να πετύχω στο τέλος, να μην μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι δική μου η μελέτη. Θέλουμε η μελέτη να θεωρηθεί ότι είναι μελέτη όλων και όλοι να πούν το είδα, το παρακολούθησα, έβλεπα κάθε μέρα τι γινότανε, είναι ανεξάρτητη μελέτη, μπορεί να μην είναι ικανοποιημένο από την έκβαση, αλλά είναι η δική μου μελέτη. Γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιος που δεν είναι ικανοποιημένο εμείς, θέλουμε ωστόσο να είναι μια μελέτη όλων των ομάδων. το αυστριακό τμήμα του Δούναβη. Είναι σχεδόν ένα υπόδειγμα. Έχει γίνει πολύ καλό συνδυασμός περιβαλλοντικών στόχων και αναγκών ναυσιπλοείας στην Αυστρία. Το Εθνικό Πάρκο από το οποίο περνάει ο Δούναβης θα σωθεί. Τα κομμάτια, το σλοβακικό και το ουγγαρέζικο τμήμα, πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι του Δούναβη. Ίσως να ξέρετε ότι ήμουν στο δικαστήριο στην Χάγη, βγήκε η απόφαση και οι δύο πλευρές βρήκαν στην απόφαση αυτό που θεωρούν καλύτερο για αυτές. Πάντα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η επίλυση του προβλήματος ωστόσο, πολιτικά τουλάχιστον, δεν είναι εύκολη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μείνω έξω από το πολιτικό, την πολιτική διάσταση. Προσπαθώ να βρω πρακτικές λύσεις. Και ίσως να τα βρούμε. Το τα τμήματα του Δούναβη στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Εκεί προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην δημιουργία συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για να αντιμετωπίζουν το ζήτημα από κοινού, διότι το το σύνορο, το είναι στο μέσο του ποταμού. Δεν μπορείς λοιπόν να, προχωρεί, να, να κάνεις ας πούμε από τη μια μεριά ε, απόφραξη και από την άλλη να μην αφήνει τίποτα. Ένα πρόβλημα στην Ρουμανία είναι το ζήτημα του οξύριγχου. Η περιοχή αυτή είναι οικότοπος του οξύριγχου και δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε τον βιότοπο αυτό. Οι προσπάθειες λοιπόν γίνονται να ώστε να κρατηθεί, να διατηρηθεί η να διατηρηθεί ο βιότοπος. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση παλεύει και πραγματικά παλεύει γιατί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπλοκη. δεν μπορούν να τα καταφέρουν εύκολα, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Θέλουμε να απλοποιήσουμε λίγο την κατάσταση, ε, στέλνοντας μια μικρή ομάδα ειδικών, λέγοντας που να κάνετε αυτό και αυτό και αυτό. Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να τους βοηθήσουμε. Αυτά είναι τα βασικότερα κομμάτια για τον Δουναβή. Σικουάνας Σκάλβης τώρα. Λιγότερα κράτη εμπλέκονται. Το βασικό πρόβλημα είναι μόνο η χρηματοδότηση. Και ο μόνος τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι εάν θέσουμε διόδια. Έχει ξεκινήσει μία διακυβερνητική ομάδα που ασχολείται με τη χρηματοδότηση, και την επιβολή διοδίων για να μειωθεί το έλλειμμα. Ένα σημείο είναι στο, στη σύνδεση αυτή, ένα σταθμό στο Τέρνχόιζεν, όπου η Φλάνδρα και η Ολλανδία ε, συζητούν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν ένα τεράστιο υδατοφράκτη που είναι ο μόνος τρόπος για να μας ε, επιτρέψει να φτάσουμε μέχρι το σκάλι, γιατί ξέρετε το λένε εσείς οικοανασχάλιδες αλλά δεν φτάνει, δεν φτάνει μέχρι το σκάλι, πραγματικά. Τσεχία τώρα. Πήγαμε στην, ε, στο, στο σημείο, στον κόβο του Ντέτσιν στον Έλβα το Μάτιο Το Ντέτσιν θα μπορούσε να συνδέσει τα γερμανικά λιμάνια με τσέχικες βιομηχανίες. Μιλήσαμε για το ενδεχόμενο κατασκευής του υδατοφράκτη εκεί. Ε, το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα ε, μεταξύ των κυβερνήσεων. Τώρα, Ιταλία, Πάδος. Εδώ διαπιστώσαμε κάτι σημαντικό. Δεν ζήτησαν χρηματοδότηση ήθελαν την υποστήριξή μας, τους την δώσαμε με, χαρά γιατί έκαναν μόνοι τους τη δουλειά. Στην ουσία τι κάνουν, ε, αναβαθμίζουν τις, ε, τα κανάλια του ΠΟ μέχρι την Μάντοβα και την Κρεμόνα για σκάφη κατηγορίας 8. Ε, κατηγορίας Α, συγγνώμη έχουν κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά και χωρίς χρηματοδότηση. Η αρχή, η λιμένος ε, Βενετίας, ο Πάολο, ο αγαπητός μας Πάολο βέβαια, αγόρασε πέντε φωτιγίδες που λειτουργούν ιονή λεωφορεία στις μεταφορές. Η η υπηρεσία αυτή ξεκίνησε σε τακτική γραμμή το Φεβρουάριο του 2009 και επαναλαμβάνω χωρίς χρηματοδότηση. Αυτά τα ειδικά. Μέχρι εδώ και να απαντήσω, αν θέλετε, σε ερωτήσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Μόνο δύο αγορητές μετά ανέφερε ε, το Δούναβι, τη Βιέννα και την Αυστρία κυρία Λίχτεμπεργκ. Ε, θέλει να παρέμβει, αλλά είμαι σίγουρος ότι η λεκάνη του Δούναβι η Επιτροπή τη υιοθέτησε. Υιοθέτησε σαν αγαπημένο της ποταμό. αυτή η Επιτροπή του Δούναβι. Όλοι αγαπούν τον Δούναβι και τη λεκάνη του Δούναβι. Η κυρία Τικάου είναι στον κατάλογο και μάλλον με τα χαρά θα αναφερθεί στην λεκάνη του Δούναβη. Και ίσως πρέπει να πάμε ακόμα πιο μακριά στον αφορά τις ε, εκτάσεις του Σικουάνα. Θα φτάσει μακριά τελικά. Λοιπόν, ο κύριος Γκρός έχει το λόγο πρώτα απ' όλα, μέρος του ΕΛΚ. Έχουμε χρόνο αλλά αυτό μην το εκλάβετε ως ε, δικαιολογία για να μακρηγορείτε. Σας ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομος. Θέλω να καλωσορίσω θερμά την πρώην συνάδελφό μας που είναι τώρα συντονίστρια και θα ήθελα να την ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνει που δεν είναι και πολύ εύκολη. Και έχουμε μια συντονίστρια που γνωρίζει το πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο, έχει θητεία σαν Υπουργός Μεταφορών, ξέρει πώς ήταν τα πράγματα, ξέρει λοιπόν και τα θέματα καλύτερα βέβαια που αφορούν την Ολλανδία και τη Φλάνδρα, γίνατε γνωστή ως ρεαλίστρια. Λοιπόν, έχω μια πολύ ρεαλιστική ερώτηση σας. Αξίζει τον κόπο να ξοδεύουν τόσα χρήματα για αυτό ή ο Ρήνος είναι η μόνη δίωδος οδός ναυσιπλοείας που αξίζει επενδύσεις διότι μπορούν να αποσβεστούν αυτές μακροχρόνια. Ε, εάν δεν είχα θέσει το ερώτημα εγώ, ο κύριος διοτι μπορουν να αποσβεστουν αυτες μακροχρονια εαν δεν σίγουρα θα το είχε θέσει. Εγώ δεν έχω πνευματική διοκτησία επί του ερωτήματος. Θέλω να ακούσω λοιπόν τη ρεαλιστική σας απάντηση αφού θεωρείστε ρεαλίστρια. Δεύτερον, Χρειάζεται συντονισμός. Έχουμε συμφωνία μεταξύ των Υπουργών Περιβάλλοντος, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι αυτά που αφορούν το περιβάλλον και τις ε, οδούς εσωτερικής ε, ναυσιπλοείας. Έχουμε και το Natura 2000 και θέλουμε να αποφύγουμε κάποια πράγματα και θέλουμε να συνεργαστούμε με αυτούς τους ανθρώπους που κατοικούν κοντά στις όχθες αυτών των ε, οδών εσωτερικής ναυσιπλοείας. Χρειάζεται συντονισμός των προσπαθειών. Χρειάζεται συντονισμός μεταξύ επαρχιών, ε, κομιτιών, αν θέλετε, επαρχιών, περιφερειών, σε χαμηλότερο επίπεδο από σε επίπεδο χωρών. Είπατε ότι χρειάζεται πρόληψη των προβλημάτων. Δεν είπατε περισσότερο, δεν αναφερθήκατε εκτενώς. Υπάρχει και το πρόβλημα ελλείψεως πόρων. Με κάποια προγράμματα μπορεί να δει κανείς ότι ότι όταν το πρόγραμμα έχει ευρωπαϊκή διάσταση, μία χώρα δίνει τα περισσότερα χρήματα. Υπάρχει αλληλεγγύη οικονομική τελικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα διάφορα συμφέροντα και δεν πρέπει να, να αργήσουμε να βρούμε λύση, γιατί υπάρχουν συμφέροντα που συγκρούνται. Ευχαριστώ για τη συντομία σας. Η κυρία Τικάο, που πιθανότατα θα δώσει απάντηση στο ερώτημα, δηλαδή κατά πόσο ο Ρήνος μόνο θα έπρεπε να πάρει χρήματα. Η κυρία Τικάο, ή μάλλον η κυρία Τσίκαο. Λοιπόν, μισό λεπτό, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, έγινε η παρουσίαση. Όπως είπε ο πρόεδρος μας, ε, εμείς αγαπάμε το Δούναβι, έχουμε υιοθετήσει το Δούναβι, η Επιτροπή μας. Do you have translation? Yeah, I had translation. Yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah, course. Uh, încă de acum 2 ani uh, am uh, încercat... Λοιπόν, πριν από δύο χρόνια περίπου προσπαθήσαμε να εισαγάγουμε στην ημερήσια διάταξη, στο πρόγραμμα της Επιτροπής Μεταφορών, αυτό το θέμα, το ώστε η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού της προηγούμενης θετίας και αυτή το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο πέρσι, ετοίμασε μια αντιπροσωπεία που πήγε Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουμανία. Θέμα της αντιπροσωπείας ήταν ο Δούναβης. Το βασικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε μετά την επίσκεψη ήταν ότι έπρεπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημιουργήσουμε μια διακομματική ομάδα για την πρόθεση του Δούναβη και αυτό είναι κάτι που θα υλοποιηθεί στις αρχές αυτής της θητείας. Ξέρουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται σχετικά στρατηγική που αφορά τη λεκάνη του Δούναβη. Να, θέλει να ασχοληθεί με θέματα μεταφορά, περιφερειακής ανάπτυξης, περιβάλλοντος, διότι ε, ε, είναι μια κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ευρωπαϊκή αξία ο Δούναβης. Για να απαντήσω στον κύριο Γκρός, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ένα θαλάσσιο αυτοκινητόδρομο που θα πηγαίνει από τη Βόρεια Θάλασσα στον Εύξηνο Πόντο και αυτό εξαρτάται από εμά. Από εμά εξαρτάται να το υλοποιήσουμε αυτό θα συντομεύσουμε κατά χιλιόμετρα την απόσταση μεταξύ βόρειας θάλασσας και ευξήνου πόντου και μπορούμε να δημιουργήσουμε διαδρόμους ε, οι οποίοι θα συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών στην Ευρώπη. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, Πώς θα συμμετάσχετε στην εκτέλεση της μελλοντικής αυτής στρατηγικής για την ανάπτυξη της λεκάνης του Δούναβη. Ξέρουμε ότι δυστυχώς όσον αφορά τις ποτάμιες μεταφορές ότι υπάρχουν κάποια τμήματα όπου υπάρχουν προβλήματα σύγκρουσης των συμφερόντων των περιβαλλοντικών και των συμφερόντων των μεταφορών. Και τι γίνεται με το δέλτα του Δουναβή, με τη διάβλο Διστροΐα η οποία είναι σημαντικό στοιχείο αυτού του διαδρόμου. Όσον αφορά το πρόγραμμα Ναϊάδες, δυστυχώς υπάρχουν χώρες, τουλάχιστον νέες χώρες, νέα κράτη-μέλη που έχουν πρόσβαση σε πολύ λίγες δυνατότητες από αυτές που προσφέρει το πρόγραμμα Ναϊάδες. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα. Ίσως μαζί μπορούμε να προετοιμάσουμε μελλοντική δράση για, την πρόσβαση, για τη βελτίωση της πρόσβασης και χρήσεως αυτού του μέσου. Σας διαβεβαιώ ότι είμαστε συνεργάτες σας, εταίροι σας και μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη των μεταφορών μέσω του Δούναβη και θέλουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη της λεκάνης του Δουναβία. Ε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στέρξ. Μετά θα δοθούν απαντήσεις στα τρία ερωτήματα και μετά θα ακολουθήσει η κυρία Λίχτεμπεργκ, κύριος Βαντάλεν και ο κύριος Κρέιμερ. Ο Ντέρκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητή Κάρλα για τις εξηγήσεις που μας έδωσες. Θεωρώ ότι αυτά που είπες ήταν πολύ θετικά. Είναι καλές ειδήσει για το πρόγραμμά σου, διότι είπε συγκεκριμένα πράγματα. Ήδη υπάρχει μεγάλη ροή εμπορευμάτων που καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα αυτής της ε, διαδρομής. Καταρχάς, αναφέρθηκες η ίδια σε συγκεκριμένα προβλήματα. Για την εμβάθυνση της ΚΙΤΙΣ ε, νομίζεις ότι υπάρχει θετική αντιμετώπιση του δυτικού κλάδου του Σκάρδη. Λοιπόν, Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν, τι ποτάμιες οδούς. Ίσως για να ρυθμίσουμε τα πράγματα θα μπορούσαμε να βάλουμε διόδια. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Ως... Φτάνουμε λοιπόν στο Σκάρβι, ήδη στη Γάνδη. Είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι θέλετε να φτάσετε μέχρι το Τέρνιους, διότι όλη η διαδρομή από τη Γάνδη μέχρι το Τέρνιους ε, είναι πιο σύντομη οδός για την μεταφόρτωση εμπορευμάτων. Μεταφόρτωση από ποντοπόρα σκάφη σε σκάφη σε ποταμόπλια. Εάν γίνει αυτό λοιπόν θα είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Εκ μέρους του κυρίου Καντράουι έχω ένα ερώτημα που κατάγεται από είναι γείτονά θέλετε, από πλευρά καταγωγή. Στην έκθεσή σα δεν αναφέρεται φράκτη, είπατε. Για μεγάλο υδατοφράκτη. Η Γάνδη είναι σημαντικό λιμάνι. Και θα πρέπει όμως σκεφτούμε τι γίνεται με τα μεγάλα πλοία όταν μιλάμε για περίπλοκους υδατοφράκτες στο Τερνούς, πρέπει να λάβουμε υπόψη και την παράκτεια, στο σχετισμό παράκτειας ακτοπλοείας και εσωτερικής ναυσιπλοείας. Λοιπόν, αυτό, αυτή την πτυχή, τη διασύνδεση, θα ήθελα να τη συμπεριλάβετε στην έκθεσή σας. Άκουσα διάφορα από αυτά που είπατε. Διαπίστωσα λοιπόν ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές ανησυχίες και ανησυχίες του τομέα των μεταφορών και καμιά φορά δεν συμφιλιώνονται οι δύο πλευρές. Συζητήσαμε εκτενώς την πολιτική για τα λιμάνια. Και εκεί μιλήσαμε για τη διασύνδεση κρατικών ενισχύσεων και των ιδιών περικολογικών μέτρων πρέπει να γίνει κάποια πρόταση για τα λιμάνια και τους εσωτερικούς λιμένες στα ποτάμια. Τι σκεφτόσαστε λοιπόν πάνω σε αυτό. Τέλος, κρίση στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ άσχημα στον τομέα για την ώρα. Σας ανησυχεί αυτό. Είναι κάτι που είναι εκτός των αρμοδιοτήτων σας. Ευχαριστώ, Ντέρκ. Θε Κάρλα να απαντήσει πρώτα στα τρία ερωτήματα και μετά επανερχόμαστε σε ένα δεύτερο γύρο. Κοιτάξτε. Αναφέρθηκαν πολλά θέματα. Ο Δούναβης είναι ένα ποτάμι κοντά στο οποίο ζουν πολλοί άνθρωποι. Συνδέει πολλές χώρες, πολλές περιοχές. Οι οποίε διασυνδέονται μεταξύ τους με αυτόν τον τόσο ωραίο ποταμό. Είμαι πεπισμένη λοιπόν ότι ασφαλώς και χρειάζεται και αξίζει τον κόπο. Έχουμε μεγάλα προβλήματα βέβαια. Πιστεύω ότι πρέπει να αναπτυχθεί και στις ε, επίπεδο ε, του εσωτερικού της ενδοχώρας ε, και μεταξύ κρατών αλλά και εντός ενός κράτους παράδειγμα μεταξύ κρατών Ουγγαρία και Σλοβενία μεταξύ δύο κρατών παλιό το πρόβλημα το οποίο βλέπουμε και πάλι στον 21ο αιώνα Ξέρουμε ότι δεν θα απαλλαγούμε γρήγορα από το πρόβλημα αυτό. Ε, πάντως θα πρέπει νομίζουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και στο μέλλον. Μεταξύ Σλοβακίας λοιπόν και Ουγγαρίας δεν θα επιληθεί εύκολα το πρόβλημα. Με, τα, με ρεαλιστικές λύσεις ασφαλώς θα πρέπει να δράσουμε. Την πολιτική δεν την ε, προσδιορίζουμε εμείς, την αφήνουμε στις ε, κυβερνήσεις, αλλά προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα τα οποία θέλει ο καθένας βέβαια να λύσει. Έχουμε λοιπόν τις δυσκολίες μας, αλλά θέλουμε και με ρεαλιστικό τρόπο να πείσουμε τις ε, κυβερνήσεις να βοηθήσουν. Και θέλουμε όλα τα κράτη να δουν ότι κάθε κράτος θα συμμετάσχει σε αυτό. Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι δεν θα συμμετέχει η Αυστρία επειδή συμμετέχει η Σερβία, Φερρυπίν. Γιατί εάν ε, αποκλειστεί η Αυστρία δεν έχει καμία πρόσβαση. Ε, είναι κλεισμένη μεταξύ Γερμανίας και Σερβίας η Αυστρία. Τα πάντα πρέπει να τα δούμε και όλοι πρέπει να δούμε ότι ζούμε μέσα σε μία αλυσίδα. Ξέρουμε σε τι επίπεδο κινούμαστε οι λύσει μπορεί να είναι μια πολιτική συμφωνία εδώ ή μια ε, ρεαλιστική αν θέλετε λύση κάπου αλλού. Νομίζω ότι μπορούμε με την πυθό να βρούμε λύσεις. Για τη σύγχρηματοδότηση των εθνικών κρατών. Δεν είμαι βέβαιος ότι, βέβαιη ότι κατάλαβα. Ναι, εγώ εννοούσα προγράμματα όπου το 80% της χρηματοδότησης καλύπτει 5-6 κράτη και το 80% ανήκει σε ένα κράτος μόνο. Και βέβαια θέλουμε συγχρηματοδότηση, όμως το εμπλεκόμενο κράτος είναι αυτό το οποίο προκαλεί και τις προσθέσεις δυσκολίες συνήθως ένα σύστημα που μπορεί ένα κράτος να είναι υποχρεωμένο να επενδύσει χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες ε, λύσεις, ε, τους ιδιωτοφράκτες, ε, τα 70-80 εκατομμύρια που ενδεχομένω κοστίζουν, αλλά πάντως ότι όταν η προστιθέμενη αξία από την επένδυση, που είναι, έχει ψηλό κόστος για το ένα κράτος, αλλά η προστιθέμενη αξία εμφανίζεται τελικά σε άλλο κράτος. Μα τα χρήματα δεν είναι ε, θέμα, δεν είναι πρόβλημα δηλαδή. Είναι πολλά τα χρήματα και ασφαλώς δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν είχαμε πρόβλημα δηλαδή να προχωρήσει ένα σχέδιο και να δούμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα. Άλλα προβλήματα έχουμε. Αλλά τα χρήματα δεν είναι πρόβλημα. Κυρία κάω, καλά θα προφέρω το όνομά σας. κάω. Στα αγγλικά. Θα ήταν πολύ καλή ιδέα, πιστεύω, να συνδυάσουμε τις ε, μεταφορές και τον τουρισμό. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, μεταφορές μέσω του, δυνα... του θα βοηθήσουν ασφαλώς τους ανθρώπους να έρθουν πιο κοντά. Εάν υπάρχει σύστημα διαμετακόμιση σύστημα το οποίο θα επιτρέπει να χρησιμοποιήσει κανεί το Δούναβι για να πάει από τη μια χώρα στην άλλη. Γιατί δεν απέχουμε τόσο πολύ. Εμείς άλλωστε πήγαμε από τη Βιέννη στην Πρατισλάβα ε, με πλοίο. Πολύ ωραίο ταξίδι. Και ασφαλώς θα απαλλάξει τους αυτοκινητοδρόμους από το, το, κυκλοφοριακό, από την επιβάρυνση στην κυκλοφοριακή. Πολύ καλή ιδέα σας και την ε, προάγουμε κι εμείς. Είναι λοιπόν ε, ήδη επιτυχημένη επιχειρημένο το εγχείρημα. Θα επιτύχει ακόμη περισσότερο πιστεύω. Intergroup, ναι, καμιά αντίρρηση. Πολύ ευχαρίστω. Στο Συμβούλιο όμως, σε ομάδα του Συμβουλίου στη Σουηδία, ο κύριος Μπίσλι, αν δεν απατώμε, πρώην συνάδελφος, μας έλεγε ε, μια ιδέα για μια intergroup και πρέπει να πω ότι <laughs> ζήλεψα κι εγώ, έλεγα μακάρι να έχω κι εγώ μια intergroup για το Δούναβε. Μακάρι. Και για τον κύριο Γκρός νομίζω ότι την απάντηση τη δίνετε εσείς. το να ε, συνδεθεί η βόρεια με τη θάλασσα, αν και δεν νομίζω ότι θα είναι πολλά τα εμπορεύματα που θα μεταφερθούν από το Ρότερνταμ ε, στην Κωνσταντζα, μάλλον προς τα έξω είναι η κίνηση στους λιμένες αυτούς και όχι προς τα μέσα. Αλλά πάντως μπορεί να περιμένει κανείς ε, μετακίνηση μεγάλων φορτίων από το Ρότερνταμ, μεγάλων όγκων φορτίων από το Ρότερνταμ στη Βιέννη ή σε κάποιο λιμένα της ε, Γερμανίας ή της Ουγγαρίας. Τεράστια απόσταση. Εάν αυτό το φορτίο φύγει από τους αυτοκινητοδρόμους που είναι τόσο επιβαρημένοι στην περιοχή αυτή, εγώ θυμάμαι πόσο πολύ δυσκολευόμουν όταν ήμουν υπουργό των μεταφορών με το Wochenende με την απαγόρευση δηλαδή κυκλοφορία των φορτηγών στους αυτοκινητοδρόμους της Βαβαρίας με την βαβαρική κυβέρνηση πόσες δυσκολίες είχαμε τα Σαββατοκύριακα ήταν απαγορευμένη κίνηση των φορτηγών μας έλεγαν όμως από τη Βαβαρία δεν αντέχουμε άλλο, δεν έχουμε άλλο περιθώριο για κίνηση φορτηγών ή άλλων αυτοκινήτων, εν πάση περιπτώσει, στους αυτοκινητοδρόμους μας. Πολύ θα βοηθήσει λοιπόν αυτό. Και αν αυτή η κίνηση πάει κατά τρόπο περιβαλλοντικά ε, σωστό οικολογικό δηλαδή, με δίκτυα ασφαλείας, με δίκτυ ασφάλειας ε, αφενός και με δίκτυ ε, προστασίας της κυκλοφορίας αφετέρου ε, με τα μέτρα εκείνα που θα αποτρέψουν την ανάπτυξη κάποιας πυρκαγιάς ή κάποιου θαλάσσιου ατυχήματος, στον, ατυχήματος στα νερά του Δούναβη. Ε, τότε ναι μπορούμε να επιτύχουμε πάρα πολλά. Και βεβαίω θα ήθελα και εγώ στο μέλλον να συμμετάσχω στην ανάπτυξη κάποια στρατηγική. Όταν ήμασταν στη Σουηδία, ήμουν εκεί για την πολιτική και τη βαλτική θάλασσα, που θεωρείται μακρό η βαλτική. Και θέλουν την αντίληψη αυτή να την εφαρμόσουν και για το Δούναβι που παρουσιάζει χαρακτηριστικά αντίστοιχα με τις Βαλτική. δηλαδη Δηλαδή περνάει μέσα από πολλά διαφορετικά κράτη-μέλη. Έχει μήκος 2.800 ε, χιλιόμετρα. Φανταστείτε έναν ε, αυτοκινητόδρομο πάνω στον οποίο ε, αντί για αυτοκίνητα κυλάν καράβια. Δεν ξέρω αν ενοχλούν αυτά που λέω τον κύριο Γκραμ ε, έτσι όπως τα περιγράφω, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η, η ιδέα που βλέπω εγώ και η ιδέα της μακροπεριφέρειας είναι νομίζω ενδιαφέρουσα γιατί συνεπάγεται μια ολιστική προσέγγιση και δεν θα επιτρέψει κάποιο να ασχοληθεί μόνο με μία πτυχή φερρυπίνη των μεταφορών ή μόνο το, για το περιβάλλον ε, να ληφθεί μέρημνα. Όχι, θα λαμβάνεται μέρημνα ολιστικά για όλου του τομεί και για τον τουρισμό και για την ανάπτυξη των παρόχθιων ε, περιοχών. Όλα αυτά τα οποία μπορεί κανείς να σκεφτεί εν ώψη της ανάπτυξης ε, μια τέτοια πλούτου. Α, νόμιζα ότι έχετε περιθώριο χρονικό μεγάλο. Όχι, όχι, μπορώ να συνεχίσω κι άλλο να μιλάω. Για την πιστορία μην με ρωτήσετε, δεν ξέρω. Δεν, μπορώ να απαντήσω, είναι πολιτικό πρόβλημα. Μας έχει ζητηθεί να μην το εγγύξουμε. Είναι ένα ζήτημα καυτό μεταξύ των κυβέρνησεων τη περιοχή και δεν θέλω εγώ να εμπλακώ. Ίσως εάν θέλετε να μου πείτε διμερώς στη συνέχεια ποια είναι τα κράτη τα οποία έχουν προβλήματα πρόσβασης συγκεκριμένα. Για τον κύριο Στέρξ. Για τον Έσκο, ε, τον ποταμό Σχέλντε. Σχέλδη. Είναι όντω περίπλοκα τα προβλήματα. Το γνωρίζετε και εσείς όπως και εγώ. Υπάρχει ένα κείμενο του 1839 συμφωνία μεταξύ Βελγίου και κάτω χωρών. Ίσως είναι λίγο απειρχιωμένα αυτά που θα σας πω λοιπόν, σωστά έχει ξεπεράσει η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει όμως γνωρίζετε για τι πράγμα μιλάω. Για δε τα διόδια, ναι ασφαλώς είναι πολύ σημαντικό θέμα. πολλά τα χρήματα και βέβαια είναι καλό ένα κανάλι καινούριο να προσφέρει και έσοδα αν θέλετε. Οι Γάλλοι είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν περισσότερο να αναπτύξουν το διαλειτουργικό ε, τομέα, δηλαδή και για τον τουρισμό και για την διαχείριση των υδάτων της περιοχής. Θέλουν να καλύψουν δηλαδή ε, με αυτή τη λύση όλους τους τομείς και προφανώς πρόκειται για ένα μεγαλειώδες έργο, εάν ε, προχωρήσει. Το Τέρνιο Εζέν θα ήταν η ταχύτερη ε, πρόσβαση για τον Σκάλδη αν και δεν είναι εύκολο πάντοτε να συνδυάζονται μεταφορές, ε, οικολογική προσέγγιση κτλ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε πάντως. Για να βοηθήσουμε τις κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίε και προσπαθούμε να αναπτύξουμε ε, προσεγγίσεις πιο ευέλικτες χωρίς όμως και να προκαλέσουμε ζημιά στο περιβάλλον. Ασφαλώς θα τηρηθεί κάθε νόμος και νομοθεσία και ασφαλώς θα προσφέρουμε και εμείς την αρρωγή μας στις κυβερνήσεις έτσι ώστε να κάνουν σεβαστή την νομοθεσία. Στις μεταφορές έχουμε πολλές δυσκολίες. Εμείς ξέρετε στις κάτω χώρες δεν έχουμε επιδοτήσεις κρατικές ενώ έχουμε να κάνουμε εδώ με τομέα στον οποίο έχουν τεράστια συμφέροντα οι στόλοι μα, ο Ολλανδικός και ο Βελγικό. Και πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε τα μέτρα που θα εισαγάγουμε να μην έχουν σαν αποτέλεσμα να φτιάξουμε πολύ ωραίε πλωτέ οδού, αλλά να μην έχει μείνει στο τέλο κανένα ε, που να μπορεί να βάλει το πλοίο του να πλεύσει. Ο πρόεδρο. Ξέρετε ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο, μέχρι τι 5 δυνατόν έχουμε ολοκληρώσει. Πέρκερ, Κλέλτσερ, Κρέμερ. Σας παρακαλώ πολύ σύντομα. Κυρία Λιχτενμπέρκερ. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση, για την παρουσίαση. Ασφαλώς έχω και εγώ τις παρατηρήσεις μου. Και ιδίω για το γεγονός ότι τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά ο Δούναβης ε, έχει άλλο πρόβλημα. Είναι οι διαφορετικές δομές, είναι άλλη δομή, όχι το, το βάθος ή το εύρος του ποταμού. Όταν πήγαμε εμείς με την αντιπροσωπεία μας, είδαμε ότι το πρόβλημα, το τεράστιο πρόβλημα, είναι ένα και μοναδικό. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει διασύνθεση μεταξύ οδικών ή σιδηροδρομικών αρτηριών και ποταμού. Ή όταν υπάρχουν δεν λειτουργούν. Είδαμε κάποιους λιμένες πάνω στο, ποτάμι που δεν, ήταν, που δεν λειτουργούσαν να κλειστεί. Η διασύνδεση, η διασύνδεση μεταξύ σιδηροδρόμου και ποταμού. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κέριο πρόβλημα στον Δούναβη. Δεν έχει ακόμα γίνει ανάλυση του ποια θα ήταν τα καταλληλότερα μέσα μεταφορών για το Δούναβη. Αν θα πρέπει να κοιτάξουμε και προς το μέλλον και να δούμε ενδεχομένω τη μεταφορά πετρελαίου από τη Μαύρη Θάλασσα μέσω του Δουνάβεως. Αν και θα αμφισβητούσα εγώ το κατά πόσο αυτό θα ήταν ο καταλληλότερος τρόπο για να μεταφερθεί το πετρέλαιο από τη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πιο σημαντικό είναι ότι από την εποχή όλων αυτών των γιουγκοσλαβικών πολέμων που ζήσαμε έχουν διαλυθεί οι διασυνδέσεις προς τον ποταμό. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν είναι κατάλληλο ο ποταμός, αρκετά ευρύς ή αρκετά βαθύ. Είναι ότι δεν έχουμε τη διασύνδεση. Η αρκετα βαθυς ειναι οτι είναι αυτή που μα λείπει ή τα σημεία μεταμφόρτωσης, ε, μετάβασης αν θέλετε. Ε, αυτό είναι που δεν βλέπουμε. Επίσης μιλήσατε για το αυστριακό σχέδιο ανατολικά της Βιέννης, ότι είναι καλύτερη ε, πρακτική, υπόδειγμα καλύτερης πρακτικής. Το αμφισβητώ αυτό. Θα έπρεπε ίσως να έχετε συνομιλήσει με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις οι οποίες είχαν εμπλακεί στην υπόθεση αυτή εξ αρχής και να κοιτάξετε με διαφορετική ματιά την υπόθεση αυτή. Το ίδιο ισχύει και για το Φιλτσχόφεν που ακούστηκε νωρίτερα. Και πάλι, πρόβλημα δεν είναι ο ποταμός, αλλά η διασύνδεση. Ο Δούναβης μπορεί να είναι πρόσφορος και για τον τουρισμό και για τις μεταφορές, εφόσον γίνεται σεβαστή η φύση. Δεν μπορούμε να καταστρέψουμε τον ποταμό και μετά να περιμένουμε την αθρώα προσέλευση των τουριστών. Ασφαλώς και ο τουρισμό προκαλεί κάποια ζημιά ή κάποια παραβίαση στη φύση, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Και φαντάζομαι ότι ο Δούναβης μπορεί να αποτελέσει το καλύτερο παράδειγμα να προσαρμοστεί το σκάφος στον ποταμό και όχι ο ποταμό στα σκάφη. Γι' αυτό θα ήθελα να σα παρακαλέσω αυτή την ιδέα το σκάφος προσαρμόσης στον ποταμό και όχι ο ποταμός στο σκάφος, να αντικαταστήσετε κέρια, κύρια ιδέα του σχεδίου σας. Λοιπόν, θα πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα. Συνδέεται, λοιπόν, δύο μεγάλες θάλασσες, τον Εύξηνο Πόντο και τη Βόρεια Θάλασσα, Ανατολική με Δυτική Ευρώπη και αυτό είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκό θέμα. Συζητείτε όμως το θέμα των υποδομών το θέμα επίσης του περιβάλλοντος, υπάρχουν ανησυχίες για το περιβάλλον. Δεν θα πρέπει να μολύνουμε, βλέπετε, τον ποταμό περισσότερο. Δεν πρέπει να συζητάμε το αν το αυγό έκανε την κότα ή η κότα το αυγό. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον διάβλο και να προωθήσουμε τις ποτάμιες μεταφορές. Είναι σημαντικό αυτό, είναι ασφαλείς οι μεταφορές σχετικά ασφαλείς μεταφορές και φιλικές προς το περιβάλλον. Δεν χρειαζόμαστε σύγκρουση μεταξύ περιβάλλοντος και υποδομών. Αν δείτε αυτό το κανάλι στο Δούναβι βλέπετε ότι υπάρχει, ε, γίνεται το έργο και δεν βλάπτουμε το περιβάλλον. Αυτοί που πανικοβάλλονται λοιπόν και φοβούνται το περιβάλλον θα πρέπει να σταματήσουν. Υπάρχει δυνατότητα συμβίωσης η σωστή υποδομή με το περιβάλλον. Αναφερθήκατε σε μια ομάδα ελέγχου. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Διάβασα σε κάποια γερμανική εφημερίδα ότι συζητείται το θέμα των μελών της ομάδας ότι γίνεται μάχη μεταξύ Μονάχου και Βερολίνου όσον αφορά το ποιος θα συμμετέχει στην ομάδα. Ερώτημα. Ξεκίνησε η ομάδα ή εξακολουθούν οι τσακωμοί. Δεύτερον, ελπίζω όπως και εσείς ότι τα αποτελέσματα της μελέτης θα είναι δεσμευτικά για όλους. Διότι αυτή η χρυσή λεωφόρος από τη Βόρεια Θάλασσα στον Ξινοπόντο θα πρέπει να έχει τύχη. Ευχαριστώ κύριε Κάντσιν. Ευχαριστώ. Είσαστε πάρα πολύ άριστοι στην παρουσίαση σας και είσαστε εκφράσατε σαφέστατες ιδέες και μας εξασφαλίσατε, μας διαβεβαιώσατε ότι δεν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Αυτό μας καθησύχασε κάπως. Αυτός ο διάδρομος που μιλάμε, αυτός ο αυτοκινητόδρομος δεν εντάσσεται στις έξι, στους έξι διαδρόμους που θεωρούμε ότι έχουν προτεραιότητα. Και το ερώτημά μου είναι αυτό. Χρονοδιάγραμμα. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα διότι δεν είναι σαν κατεπήγον ζήτημα αυτό ανάμεσα στους έξι στόχους προτεραιότητας. Πώς συνδυάζεται η μεταφορά η θαλάσσια με την ποτάμια. Είναι πολύ σημαντική η διασύνδεση, κυρίως αν όπως λέγατε Λάβω υπόψη τα όσα είπε ο πρώην συνάδελφος Κώστα, ο κ. Κώστα που ασχολήθηκε με τον Πάδο. Το πρώτο κομμάτι ρυθμίστηκε. Υπάρχουν οι δυνατότητες ε, να μπορούμε να κάνουμε κάτι για να λάβουμε υπόψη και το ενεργειακό θέμα. Και αυτό συνδέεται με το θαλάσσιο κομμάτι. Όταν συζητούσαν πλέον τα, την Τεργέστη, τη Ραβένα, τη Βενετία, τα λιμάνια, τα θαλάσσια της Αδριατικής. Λοιπόν, και λίγο για την αυσιπλοεία στον Πάδο. Αυτό το πρόγραμμα θα, θα ενταχθεί σε ένα πλαίσιο, θα είναι ολοκληρωμένο. Αυτά θα ήθελα να ρωτήσω. Τελικός ομιλητής, ο κ. Κρέιμερ. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σαφείς να μιλάμε στα ράτα. Το 80% των πλωτών μεταφορών περνάνε από τον ε, δούναβη στην ε, Ευρώπη. Πολύ καλά λοιπόν να το συνδέσουμε με τη Βόρεια Θάλασσα. Τα υπόλοιπα είναι αυτά τα οποία θα χρειαστούν υποστήριξη χρηματοδότηση δηλαδή γιατί δεν υπάρχουν αρκετές ε, διασυνδέσεις, γιατί δεν υπάρχει αρκετή κίνηση και γιατί εξαρτώμαστε πάρα πολύ από τις, καιρικέ συνθήκες. Στον Έλβε παραδείγματι στη Γερμανία έχουμε από το Βερολίνο στο Ανόβερο φτιάξει μία δίωδο για ένα πλοίο που περνάει όχι μια φορά την ώρα, ούτε μια φορά την ημέρα, μια φορά την εβδομάδα. Υπάρχει λοιπόν διασύνδεση, έχει γίνει η δουλειά, θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε, αλλά δεν παίρνουν να περάσει το τεράστιο σκάφο. Κι εγώ. Από το Ίγκεστατ στην Μαύρη Θάλασσα που πήγα και ταξίδεψα. Ναι, πολύ ωραία. Υπάρχουν και τα πλοία που θα σα κατεβάσουν έτσι. Αλλά όπω και στο παρελθόν <laughs> και στο παρελθόν λέγαμε από τον ε, Ρήνο στο Δούναβι ε, ship ahoy. Τώρα λέμε ahoy. Πού είναι το καράβι. Γι' αυτό λοιπόν, ε, όχι, όχι, μην Έτσι είναι η κατάσταση. Δεν περνάνε πλέον τα σκάφη. Υπαρξιακά, ναι, μπορεί να υπάρχει ζήτημα διασύνδεση, αλλά το 80% περνάει από το Δούναβι. Το υπόλοιπο 20% τι κάνει τώρα από τη Βαλτική μέχρι την ε, Μαύρη Θάλασσα, αν θέλετε να βάλετε τεράστια σκάφη και πρέπει να γίνει η διάνοιξη και δεν ξέρω τι, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό. Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη δε, γιατί ήμουνα σε μια συζήτηση που ε, ρώτησα πόσα χρήματα νομίζω σας προσφέρει χρηματοδοτώντας η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστο 80-85% ήταν η απάντηση. Ναι γιατί μην ξεχνάμε ότι και στι χώρε τουλάχιστον για τη Γερμανία που ξέρω και μπορώ να μιλάω, η ε, κατασκευαστική πολιτική, για να μην πω η κατασκευαστική μαφία, είναι εκείνη που καθορίζει και τις επιλογές. Και Αντίστοιχα για τα, μέσα των, για τα κονδύλια που διατίθεται για τις μεταφορές. Από την άλλη όταν έχουμε μόνο ένα-δύο πλοία, ίσω είναι ακραία η απέτηση της χρηματοδότησης όταν μάλιστα είναι τόσο χαμηλή η λυπή επιβάρυνση οικονομική για, τα, για τις πλωτές αυτές οδούς. Και αν θέλουμε να αναπτύξουμε τον Δούναβη, τον τουρισμό καλύτερα στον Δούναβη, ας ξεχάσουμε οποιαδήποτε ανάπτυξη τουρισμού ή αν αρχίσουν να περνάνε μεγάλα σκάφη από τον Δούναβη. Ας μην προσαρμόσουμε λοιπόν τον ποταμό στα καράβια, αλλά τα καράβια στον ποταμό με συγχωρείτε που μίλησα έτσι σταράτα, γιατί μια και ακούστηκε το όνομά μου νωρίτερα, θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρη η εικόνα, δεν είναι δυνατόν να τα αποσιωπούμε όλα αυτά. Σα είπα, ε, κανάλι, Δούνα, ε, κανάλι Βερολίνο Ανόβερο, κάθε τόσο ακυρώνεται και κάποιο έργο διότι δεν υπάρχει καθόλου κίνηση. Το μόνο που γίνεται σε αυτήν την περίπτωση με, τις νέα, με τα νέα σχέδια κτλ. είναι να εξασφαλίσουν κάποιε θέσει εργασία. Είδε τι, τι κάνατε. Αρχίζουν διάφοροι και θέλουν το λόγο. Ναι, πολύ σύντομα. Αυτό, α, αυτή η τοποθέτηση υποτίθεται ότι ήταν ερώτηση, έτσι. Μα ήθελα να σου απαντήσω. Λοιπόν, εμάς Μάικ, μας αρέσει ο Δούναβης, δεν το κατάλαβες αυτό. Κάραλα να απαντήσεις. προς την κυρία προς την κυρία Λίχτενμπεργκερ και όχι Στάινμπεργκερ. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Χωρίς συνδέσεις δεν υπάρχει ναυσιπλοεία. και χωρίς ναυσιπλοεία δεν υπάρχουν λιμένε. αλλά όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε παράλληλα και όχι το ένα μετά το άλλο. Μπορεί να έχουμε ένα λιμάνι, ένα ποταμό, συγγνώμη, αλλά αν δεν έχουμε σημεία μετεπιβίβαση, δεν είναι χρήσιμο το ποτάμι. Εξού και η σημασία του να δουλεύουμε για την διασυνδεσιμότητα των ε, μέσων, για, τα για την χρήση από κοινού μέσων μεταφοράς στο σύνολο. Σε ό,τι αφορά την ανάλυση του είδους των εμπορευμάτων, θα σας απαντούσα το εξής, ότι οι συνδέσεις πρέπει να γίνουν από τις κυβερνήσεις των παραδουνάβιων χωρών. Δηλαδή, από το εργοστάσιο στο λιμάνι. Και αυτό θα μας γλιτώσει πολύ αυτοκινητόδρομο, αυτό είναι σίγουρο. Ξέρετε, εγώ είμαι Ολλανδί και πραγματικά στην Ολλανδία αν δεν είχαμε εσωτερικές πρωτέ οδού, δεν θα ξέραμε τι να κάνουμε αν δεν μπορούσαμε να περάσουμε τα πρώτα εμπορεύματά μας από το ποτάμι. λέτε κύριε Κράμερ ότι δεν μπαίνουν μεγάλα πλοία, ελάτε στο σπίτι μου. Στο σκάλδι πάνω μένω και εκεί θα δείτε κάτι τεράστια πλοία, κρουαζιερόπλοια που ανεβαίνουν τον ποταμό από την Κωνσταντζα που ανταγωνίζονται τα μεγάλα κοντέινερ ε, πάνε τόσο κοντά που προσπαθούν να τα δουν, να τα πιάσουν. Και πραγματικά μου κόβει την ανάσα όταν τα βλέπω. Στο δυτικό σκάλιδι υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες. Μην, μην ναι, συγκρίνουμε τον Δούναβη με το σκάλδι. Αλλά είναι δύσκολα τα και εκεί. Μπορείς λοιπόν να συνδέσεις και να συνδυάσεις μεγάλα σκάφη και τουρισμό χωρίς πρόβλημα. Τώρα, το αυστριακό σχέδιο, ο διευθυντής του εθνικού, ο διαχειριστής του έργου του, του Εθνικού Παδρυμού, με τον οποίο είχαμε μιλήσει, μας είχε πει τελείω διαφορετικά πράγματα. Τέλο πάντων, μπορεί να μιλάτε με άλλου ανθρώπου και όχι με του ίδιου με του οποίου μιλάω εγώ. Θα επανέλθω και θα του ρωτήσω. Το τελευταίο κομμάτι του ποταμού το χαρακτηρίζουν οι ντόπιοι ως ελευθέρας διέλευσης ποτάμι. Free floating. Το θέμα λοιπόν δεν είναι η επιμελητία και όταν μιλώ για επιμελητία ε, θα σας έλεγα επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή μην κοιτάτε το ποτάμι κοιτάτε την δεκάνη του ποταμού γιατί αυτό μπορεί να αφαιρέσει πάρα πολλά φωτιά από το δρόμο ο κ. Βαν είπε ότι η θαλάσσια, η μεταφορά μέσω πλωτή οδού είναι ασφαλής και χωρίς ατυχήματα. Όντως δεν υπάρχουν πολλά, σχεδόν κανένα ατύχημα στα ποτάμια. Στην Ολλανδία κανένα. Δύσκολο μπορεί να πει κάποιος ότι το κανάλι Μάιν Δουνάβεως είναι ένα πολύ εξαιρετικό υπόδειγμα γιατί δεν είναι φυσικό ε, δεν είναι φυσικός διάβλος είναι μια, ένα τεχνητό κανάλι και άρα ε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για φυσικό περιβάλλον εκεί είναι μια πολύ όμορφη σύνδεση αλλά τη σκάψουμε εμείς η ομάδα παρακολούθησης έχει ξεκινήσει να δουλεύει αλλά είναι δυσαρεστημένοι και λυπημένοι. Δεν έχουν αρκετούς για τις μεταφορές, δεν έχουν αρκετούς για το περιβάλλον. Εγώ αυτό που τους λέω είναι αντί να τσακώνεστε αρχίστε να δουλεύετε. Υπάρχει λοιπόν η ομάδα Παρακολούθησε αλλά τώρα αντί να τσακώνται πρέπει να αρχίσουν να δουλεύουν. Για τον κύριο Γκρατσιάν. Ο Πάδος. Είναι προτεραιότητα για αυτούς, γι' αυτό και το έκαναν μόνοι τους. Και έκαναν και πολύ καλή δουλειά, όπως σας είπα. Και αφαίρεσαν πολύ εμπόρευμα από τον, τις οδικές μεταφορές από το Φεβρουάριο και μετά. Ελπίζω αυτή η τάση να συνεχιστεί. Είπατε και κάτι για την ε, ένταξη, αλλά δεν το κατάλαβα στη μετάφραση. Αν, τι θέλετε, τι είπατε, τι εννοούσατε ακριβώς. Για την ένταξη, την, το συνδυασμό με τις θαλάσσιες μεταφορές που πήγαινε από τη Μάντοβα, Κρεμόνα, Βενετία και συνδεόταν με την Αδριατική, με, την, με, την, με τη θαλάσσια μεταφορά ε, από τη Βενετία και μετά. Αυτό απαιτεί ωστόσο να υπάρξει μια ε, διασύνδεση ποτάμιων και θαλάσσιων λιμένων. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, μα θα το κάνουνε, θα το κάνουνε. Το έκαναν κιόλας με την να ναυσιπλοεία έχει ήδη γίνει και τώρα υπάρχουν πολλές μεταφορές ε, φεύγει πολύ εμπόρευμα από την Πρέσα και αυτό θέλουμε να το κάνουμε ε, συνδέοντας τις υποδομές του Δουνάβεως με τις υποδομές των ρωσικών ποταμών Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα σύνδεση. Νομίζω ότι τα είπα όλα, ε. Ευχαριστώ την Κάρλα. Όλοι οι άλλοι απάντησαν σε εσά, κύριε Κρέμερ. Πώς δεν απαντήθηκε η ερώτησή σας. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει η ε, χρήση των πλωτών οδών παρά όλες τις επενδύσεις μειωθεί σημαντικά. Θα έπρεπε και οι επενδύσεις να μειωθούν αντίστοιχα εφόσον δεν χρησιμοποιούνται. Μα υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις αύξηση ίσω, αλλά γενικά στην Ευρώπη στις πλωτές μεταφορές είναι πτωτική, ραγδαία πτωτική εικόνα. Michael, θα μπορούσε να θέσει το ίδιο ερώτημα στην, ε, για τη μείωση τη, του, της δραστηριότητας του κλάδου αλλά είδαμε ότι διακόπτεται 40% των κοντέινερ στην Αμβέρσα που δεν είναι πάνω στον Ρήνο φεύγουν με πλωτή οδό με εσωτερική πλωτή οδό άρα βλέπετε ότι υπάρχουν διαφορετικέ απόψεις. Τέλο πάντων αυτό έρχεται και, εσύ και ε, επιβεβαιώνω αυτό που θέλω να πω ότι η δική σου παρέμβαση Κάρλα δημιούργησε μεγαλύτερη κινητικότητα μεταξύ των ε, βουλευτών από ότι όλες οι άλλες μαζί. Νομίζω δεν ξέρω είναι καλό ή κακό. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλό και σε συγχαίρω για τη δουλειά που κάνει, έκανες. Ευχαριστώ πολύ για την συνεισφορά και Ελπίζω να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Next up is um, Mr. on the rail Ο κύριος Τέλικα για την ε, Rail Baltica. Καθυστερήσαμε και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Το καταλαβαίνετε βέβαια. Και έχουμε και τον κύριο Βίνγκ για το ERTMS. Και ξέρω ότι δεν τζαγκώνονται για το ERTMS οι βουλευτές, οπότε δεν νομίζω να υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Κύριε Τέλικατ, έχετε το λόγο. Για την Rail Baltica. Ευχαριστώ. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Θα είμαι πολύ... Ξέρω ότι καθυστερούμε και θα περιορίσω την παρέμβασή μου. Απλά να πω ότι την τελευταία φορά που είχα έρθει εδώ δεξιά μου καθόταν ο Κάρλ Βαν Μίρτ και θέλω απλά να θυμίσω την ε, σημαντική συνεισφορά του στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Αυτή μια προσωπική εισαγωγή. Πιστεύω ότι χάσαμε έναν μεγάλο συνάδελφο, μεγάλο Ευρωπαίο και εξαιρετικό συνεργάτη. Rail Baltica τώρα. Να συνοψίσω την κατάσταση όπως είναι σήμερα. Κάτι που έγινε είναι ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια βαθιά ύφεση και η οικονομική κάμψη που έπλεξε ιδιαίτερα τις χώρες της Βαλτικής. Η μείωση του ΑΕΠ ήταν σε, ε, σε διψήφια νούμερα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο σημείο αυτό. Πρόκειται για σημαντική δυσκολία. Μπορεί να την περιγράψουμε και στις πολιτικές συζητήσεις για την περικοπή των οικονομικών, τις περικοπές στον προπολογισμό ιδιαίτερα στη Λετωνία. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε σίγουρα ότι θα υπάρξει καθυστέρηση αναμενόμενη προφανώς τώρα αλλά όχι πριν από δύο χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν να βρεθήκαμε μάλλον κατά ε, απέναντι σε σοβαρά προβλήματα. Σε κάποια σημεία υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των τεσσάρων χωρών ή των τεσσάρων συν μία όπου οι ιδιωτικοί, οι ιδιωτικοί φορείς προσπαθούν να δώσουν συγκεκριμένες λύσεις χωρίς να υπάρχει ωστόσο μείωση στη Βαλτική. Αυτό είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουμε σύντομα. Ίσως να πρέπει να περιορίσουμε τις δραστηριότητε, αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε και κάπως πιο δημιουργικοί, αναζητώντας την χρηματοδότηση και βοηθώντας και λίγο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, ε, ωστόσο αυτό είναι μια πρόσκληση ανοιχτή προς την Επιτροπή να εξετάσει θέματα όπως τη τον συνδυασμό κάποιων πηγών. Υπάρχει δέσμευση μεν, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μία επιβράδυνση που δεν νομίζω ότι θα οδηγεί σε σοβαρές ε, καθυστερήσεις στην Ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει δομέ, διαδικασίες εξυγχρονισμού στην Νότια Εστονία, στην, ε, παραμεθώ, στην παραμοθόρια περιοχή μεταξύ ε, Εσθονίας ε, και Λετωνίας, μια περιοχή που η ιστορία έχει χωρίσει την πόλη, τη διπλή πόλη Βάλγα και Βάλκα. Ταυτόχρονα εξετάζουμε το πώς θα επιταχύνουμε αλλά και με δεδομένη την οικονομική κατάσταση πώς θα μειώσουμε το κόστος του σχεδίου στη Λιθουανία εξετάζουμε προτείναμε μάλλον στην κυβέρνηση της Λιθουανίας μια σειρά εναλλακτικών λύσεων που θα περικόψουν κατά 50% σχεδόν το κόστος. Αυτό περιλαμβάνει ας πούμε την δημιουργία διπλής γραμμής ε, και να περιορίσουμε το εύρος γραμμής που είναι το ρωσικό εύρος κατά κάποια εκατοστά για να το κάνουμε το, το στάνταρ ευρωπαϊκό. υπάρχει μια ανοιχτή στάση της κυβέρνησης. Όχι των, ε, του, του οργανισμού συνδεδόμενων, αλλά τέλος πάντων. Στην ε, Λετωνία στην Πολωνία συγγνώμη, υπήρχαν μια σειρά ερωτηματικών στο παρελθόν. Το ίδιο ε, υπάρχει και τώρα. Το βασικό πρόβλημα αφορά το κομμάτι μεταξύ του Μπιάλιστοκ και της παραμεθορίου με την Λιθουανία που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ε, ολοκλήρωση του έργου. Πάντως δεν υπάρχουν αρνητικά, τελείως αρνητικές θέσεις. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι η υποστήριξη του έργου από την Φιλανδία που δείχνει ότι είναι και βιώσιμο οικονομικά. Μιλήσαμε πριν από λίγο για τα λιμάνια Πρέπει να σας πω ότι η υποστήριξη της πόλεως του Ελσίνκη στην Rail Baltica ως βασικού τμήματος ανάπτυξης περιοχής είναι μια ενδιαφέρουσα υποστήριξη. Εξίσου ενδιαφέρον είναι το πώς το καινούργιο λιμάνι του Βασάρι συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. Αν δούμε τα βασικά προβλήματα που έχουμε μπροστά μας, θα έλεγα ότι είναι τα εξής Πρώτον, θα χρειαστεί να προσαρμόσουμε το θέμα του εύρους γραμμής. Είναι και οικονομικό, αλλά η Λιθουανία που ήταν ο κινητήρας της ε, Rail Baltica όλη αυτή την περίοδο θεωρεί ότι είναι ένα ενδιαφέρον θέμα που πληρεί τις διάφορες εναλλακτικές ε, λύσεις, αλλά που αντιμετωπίζει αντί, αντιστάσεις στις χώρες. Το ζήτημα είναι πού θα μπει το κλειδί της αλλαγής ε, του εύρους γραμμής ή πού, πώς θα αντιμετωπιστούν τα, βασι... αντίστοιχα προβλήματα της, δια... της διαφοράς εύρους μεταξύ της ρωσικής γραμμής και της ευρωπαϊκής. Και το ερώτημα που μπορεί να τεθεί είναι με την υφιστάμενη κατάσταση πόσο μπορούμε να δουλέψουμε στην κατεύθυνση αυτή. Ε, θα έπρεπε ωστόσο να διασφαλίσουμε ότι οι δομές επιμελητίας που βρίσκονται μεταξύ του πολωνολιθουανικού ε, κομματιού, του, του, κομματιού στα πολωνολιθουανικά σύνορα μέχρι το Ταλίν πρέπει να αποκτήσει μια ενιαία ένα ενιαίο εύρος και αυτό δείχνει και τη σημασία του κάουνας την του κόμβου του κάουνας. Οπότε θα πρέπει να καταλάβουμε από την αντίδραση σε αυτό το ερώτημα αν το έργο είναι βιώσιμο και αν το κάουνας πρέπει να συνδεθεί με τη Βία Μπάλτικα για αυτούς τους λόγους. Και αυτό είναι από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να δούμε. Είπαμε το εύρος γραμμής στην επιλογή που υποβάλαμε στην κυβέρνηση της Λουφανίας και στις εταίρες χώρες, στις χώρες είναι ότι μπορούμε να φέρουμε μέχρι το κάουνας την, το ευρωπαϊκό εύρος γραμμής. Εγώ θα έλεγα ότι στο πλαίσιο αυτό έχουμε δυνατότητες να πετύχουμε και ταυτόχρονα απαιτούμε θα έχουμε μάλλον, όχι απαιτούμε, ζητήσαμε και θα λάβουμε από την πολωνική κυβέρνηση ε, τον σχολιασμό τους. Ένα θέμα που δεν είναι κομμάτι του Via Baltica αυτό καθεαυτό αλλά μας απασχόληση γιατί θεωρούμε ότι έχουμε μια εντολή με τον James Ποντ είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητες εμπορευματικών μεταφορών είναι ανοιχτέ στον ανταγωνισμό παντού στην περιοχή αυτή. Μπορεί αυτό θεωρητικά να είναι εύκολο, στην πράξη δεν είναι ωστόσο. Για τον απλό λόγο ότι δεν υπάρχουν δεν υπάρχει ζήτηση, αυξανόμενη ζήτηση από ιδιώτες. Υπάρχουν κάποιοι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, αυξάνεται αλλά παράλληλα με την αύξηση της, ε, του δυναμικού της γραμμής. Και βέβαια να πω ότι όταν ότι μπορεί να έχουν πολύ θετική ανταπόκριση και συνεργασία με τη Λουφανία, Φερρυπίν, με την κυβέρνηση, με το δημόσιο γενικά. Ωστόσο, η ε, διαχείριση, η διοίκηση του της εταιρείας σιδηροδρόμων ε, στην ε, Λιθουανία φαίνεται ότι καταραίει σιγά σιγά. Λοιπόν, πάντα θέλουμε συνεργασία με τους διαφόρους διαφερομένους του δρομικού τομέα που θέλουν να είναι παρόντες σε αυτό. Και αυτό είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθούμε τις επόμενες ημέρες. Κάτι που συζητήθηκε ξανά στα πλαίσια της εντολής που δόθηκε είναι το θέμα των τερματικών, των διαλειτουργικών που συνδέονται οι διάφορες μορφές μεταφορών και η διασύνδεση με, το, με τα λιμάνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, η των προγραμμάτων, η ανάπτυξη την περιφερειακή και αυτή η περιφέρεια το χρειάζεται. Αν κοιτάξετε τι γίνεται στο Κάουνας, δεν είναι μόνο θέμα αυτού της διαδρόμου της Βαλτικής. Αν δείτε το χάρτη, ε, νομίζω ότι είναι σαφές πόσο σημαντική είναι η διασύνδεση με τα λιμάνια της ε, περιοχής, είτε είναι η Ρήγα, το Κρέμπεντα, το Ταλίν. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Θα θέλαμε να έχουμε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, πολλαπλό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην προσπάθειά μας και βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς ιδιωτικών επενδυτικών στην περιοχή και για την ανάπτυξη των λιμένων. Κατά την άποψή μου νομίζω ότι αυτό θα ήθελα να το αναλάβω. Θα ήθελα αυτή η επένδυση ε, να δοθεί για στρατηγικού λόγους κυρίως από τους ενδιαφερομένους Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και πιστεύω ότι ε, το περιβάλλον θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό και θα έχουμε και ανταγωνιστές που θα έρχονται από αλλού. Η παρόδο ότι η πρόθεση των επιχειρηματιών ε, είναι κάτι που έχει σημασία για το πρόγραμμα αυτό και σε δύο εβδομάδες θα γίνει μια συνάντηση με πολιτικούς κύκλους και επιχειρηματικούς κύκλους σε μια διάσκεψη. Στο Βίλνιος θα διεξαχθεί αυτή η συνάντηση και ο αριθμός των συμμετεχόντων και από Ευρώπη και από την Ασία ε, είναι πολύ εντυπωσιακό. Ε, αυτό αποτελεί έναν από τους στόχους μας. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, όπως σας υποσχέθηκα, προσπάθησα να είμαι σύντομος λόγω χρονικών περιορισμών και άφησα αρκετά πράγματα τα οποία θα τα βρείτε στην έκθεση, αλλά θα ήθελα να συνοψίσω κλείνοντα. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε προχωρήσει σημαντικά χάρη στην νοτροπία, στη στάση και την προσπάθεια που κατεβλήθη στις χώρες αυτές το τελευταίο δωδεκάμινο. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία θα μπορούσαν να αναφερθούν και συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση. Δεύτερον, έχουμε αυξανόμενο ενδιαφέρον ακόμα και την περίοδο της ύφεση από τους ενδιαφερομένους του σιδηρομικού τομέα, τους μεταφορείς εμπορευμάτων ε, και από Ευρώπη και από Ασία. Και τα ασιατικά κεφάλαια εξετάζουν το θέμα των υποδομών των λιμένων, παρόλο που βεβαίως πλήττονται και στην Ασία εξίσου από την ύφεση. Τρίτον, θα πρέπει να σκεφτούμε ε, ποια είναι η παρούσα οικονομική κατάσταση και να δούμε όμως σε αυτά τα πλαίσια τι προσέγγιση πρέπει να ακολουθήσουμε. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να, ε, το Rail Baltica να υλοποιηθεί με χαμηλό κόστος και έκανα συγκεκριμένες προτάσεις που λαμβάνονται εδώ, κυρίως στη Λιθουανία. Εκεί μιλάμε για τις μεγαλύτερες δαπάνες όσον αφορά το Rail Baltica. Ε, θα, θα απορροφηθούν τα περισσότερα χρήματα εκεί. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε πέρα από αυτά που ήδη παρέχονται αν μπορούμε μέσω δημιουργικότητας να διευκολύνουμε τα πράγματα τον επόμενο χρόνο, τα επόμενα δύο χρόνια για εκείνε τι χώρε που έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά, όπως είναι η Λιθουανία, η Λετωνία, αλλά κυρίως ε, η Λετωνία έχει πληγεί πολύ σκληρά και μετά θα πρέπει να ασχοληθούμε με ένα θέμα που δεν είναι πολιτικό-οικονομικό, είναι στατικικό. Ε, και αυτό είναι το φάρδος των σιδηροτροχιών. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από ότι απλώς να ενταχθούν οι βαλτικές περιοχές ε, στην υπόλοιπη εσωτερική αγορά. Είναι ευαίσθητο, δύσκολο θέμα που έχει προτεραιότητα. Ε, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι καλύτερο θα ήταν να αφήσω ένα χρόνο για τα απαντήσεις. Διότι έχουμε μείνει πίσω χρονικά και η Κάρλα ήταν πολύ υπομονετική. Ο Κάρολ μάλλον, ο Κάρλ ε, είναι πολύ υπομονετικός και περιμένει να έρθει η σειρά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα και αυτό ναι, θα τον, ε, θα, θα, θα τον βάλουμε στο στόχαστρο και τον Κάρελ Βίνκ. Ο κ. Ζασάντα πρώτος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, για πρώτη φορά έχω την τιμή να πάρω το λόγο και να τοποθετηθώ εκ μέρους του ΕΛΚ και αυτό το πρόγραμμα που συζητούμε είναι πολύ σημαντικό και για την Πολωνία και τις άλλες βαλτικές χώρες είναι σημαντικό. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Μίλης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς και την ομάδα σας έξοχη δουλειά που κάνατε και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουν τα πράγματα διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο αυτό. Βασικός στόχος του Rail Baltica είναι η ανάπτυξη ποιοτικών μεταφορικών οδών που θα διασυνδέουν τις βαλτικές χώρες και την Πολωνία συμπεριλαμβανομένου και του κόμβου της Βαρσοβίας και κάλυψης και άλλων χωρών που ακολουθούν στη διαδρομή. Δεν υπάρχει αυτή η διασύνδεση και θα μπορούσε, αν γίνει, να είναι εναλλακτική λύση όσον αφορά τις οδικές μεταφορές. Και ξέρετε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στους δρόμους μας. Πόσο ε, μπλοκαρισμένοι είναι οι δρόμοι μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το ταχύτερο δυνατό να υλοποιηθεί το Rail Baltica. Για την ώρα μας οι βαλτικές χώρες δεν χρησιμοποιούν ε, τις υδρομικές μεταφορές όσον αφορά τη διαδρομή βορρά-νότου, όσον αφορά τα εμπορεύματα. Η εξυγχρονισμένη αυτή η γραμμή ελπίζουμε ότι θα αυξήσει αυτού του είδους τις μεταφορές μεταξύ βαλτικών χωρών και ε, σύνδεση με σκανδιναβικές χώρες και ιδιαίτερα με την Φιλανδία αλλά ίσως και με ασιατικές χώρες θα μπορέσουμε να συνδεθούμε καλύτερα. Ε, ένα τέτοιο σύγχρονο σιδηροδρομικό σύστημα θα βλάπτει λιγότερο το περιβάλλον, θα μειώσει τη συμφόρηση στους δρόμους και δεχομένως θα βελτιώσει και τις συνθήκες για μια μεγαλύτερη περιφερειακή ανάπτυξη των χωρών μας. Έχω κάποιες ερωτήσεις που θα ήθελα να σας θέσω. Σωστά παρατηρήσατε ότι η κρίση είναι πολύ οδυνηρή και πλήττει τις βαλτικές χώρες, όλος ιδιαίτερος, και ίσως αυτές οι χώρες να μην βλέπουν να υπάρχει ανάγκη για μεταφορικές υπηρεσίες σε αυτή τη φάση. Έχετε κάνει προσωμείωση των επιβατικών ροών κατά τη διαδρομή της Rail Baltica καθώς και την μετατόπιση από τις οδικές μεταφορές προς τις σιδηροδρομικές. Το εξετάσατε αυτό το πρόβλημα. Αν λειτουργήσει και όποτε λειτουργήσει η Rail Baltica, αναφερθήκατε επίσης στο, στην, ευρωπαϊκή, στην ευρωπαϊκή απόσταση των σιδηροτροχιών προς το Κάουνας. Είναι βιώσιμο αυτό το πρόγραμμα οικονομικά και κάτι άλλο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό τις ώρες της κρίσης, οι επενδύσεις που απαιτούνται, οι ιδιωτικές επενδύσεις επίσης, του ιδιωτικού τομέα. Βέβαια, ενέχουν κάποιους κινδύνους αυτές οι επενδύσεις. Μπορείτε να κινητοποιήσετε και να προσελκύσετε ιδιωτικά κεφάλαια. Ευχαριστώ κύριε Ζασάρ. Η κυρία Σάλισα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ για την παρουσίαση της κατάστασης. Θα μου επιτρέψετε όμως να περάσω στην εσθονική γλώσσα. Εξ όσων γνωρίζω, ο Οικονομίας και Τηλεπικοινωνιών της Εστονίας ε, και μεταφορών μάλλον της ε, Εστονίας ενδιαφέρεται για ένα σχέδιο για ε, τρένο υψηλής ταχύτητας που έχει προχωρήσει μένα αλλά ε, παρουσιάζει κάποια προβλήματα ως προς την επόμενη φάση, την μελέτη σκοπιμότητας. Ερωτώ λοιπόν, εάν δεν μπορέσει να επιβιώσει αλόβητη από τη μεγάλη οικονομική κρίση η Βαλτική. Εάν δεν μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας, έχετε κάποιες λύσεις από την Επιτροπή. Ε, στο όχι ίσως έτοιμες λύσεις, αλλά κάποιες ιδέες για την επαναχρηματοδότηση, των, για την ε, ενίσχυση της χρηματοδότησης ε, τέτοιων σχεδίων στην Βαλτική. Δεν έχουμε να κάνουμε ένα σχέδιο που θα καλύπτει πάνω από, χίλια χιλιόμετρα των διευρωπαϊκών δικτύων. Για την Εστονία. Οι κύριες οδικές αρτηρίες της Εστονίας αντιμετωπίζουν μεγάλη συμφόρηση από την αυξημένη παρουσία φορτηγών και κάθε εβδομάδα έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα λόγω των ε, της έντονης παρουσίας των φορτηγών στις ε, οδικές μας αρτηρίες. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με υψηλό κινδυνό και δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξε προς το μέλλον του εγχειρήματο αυτού. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ε, ικανοποιητικές απαντήσεις. Ευχαριστώ και τέλειο κύριος Κρέμας. Καταρχάς, θεωρώ ότι είναι συνθηκολόγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέτηση από τις προσπαθίες της, το γεγονός ότι ύστερα από πέντε χρόνια δεν έχει ακόμη καταφέρει να συμφωνήσει και να προχωρήσει. Ξέρω ότι είχατε πει σε κάποια φάση ότι μπορούμε να προχωρήσουμε για διασύνδεση με τη Ρωσία, αλλά αν αναλογιστεί κανείς ότι στις ε, μεγάλου εύρου αποφάσισε να κάνει την ε, μετατροπή της και ανέλαβε τον κίνδυνο γιατί υπήρχαν πολλά εσωτερικά προβλήματα, ε, μειονεκτήματα στη διασύνδεση πρώτα απ' όλα της Μαδρίτης με τη Σεβίλη με, με ε, ευρεία σειροτροχιά. Ε, ρωτώ λοιπόν πρώτα απ' όλα σε ποιο βαθμό έχετε προχωρήσει αυτή τη στιγμή στην μετατροπή για τις εμπορευματικές μεταφορές, τις δρομικές μεταφορές και δεύτερον για το Κάουνας υπήρχε μια υπήρχαν προβλήματα υπήρχαν ε, ίχνη ε, αν θέλετε ή μάλλον υπήρχε σιδηροτροχιά η οποία πως έπρεπε να ε, εξυγχρονιστεί όμως είναι διατεθειμένη η Πολωνία να ξυγχρονιστει ομως ειναι διατεθειμενη η πολωνια να αναπτυξει τη σιδηροτροχιά με βάση τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκές μέχρι το Κάουνας από τη δική της την πλευρά δηλαδή και μέχρι το Κάουνας θα μπορέσει να γίνει αυτό για να προχωρήσουμε λίγο ακόμα. Γιατί αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Επίσης αυτό που δεν κατάλαβα είναι που ακριβώς βρίσκονται τα προβλήματα της ε, χάραξης με την Βία Μπάλτικα και αν έχουν επιληθεί ή όχι. Και επίση όταν έχετε στην αναφορά σας 5.000, την αναφορά σε 5.000 φορτηγά την ημέρα στην ε, την περιοχή αυτή και ότι είναι το 20 πλάσιο από τις σιδηροδρομικές μεταφορές ο όγκος ε, των μεταφερομένων ε, φορτίων, ε, τότε πώς είναι δυνατόν να μου λέτε δεν, μπορεί, δεν θέλουν οι Πολωνοί και δεν μπορούν οι Λιθουανοί ή θέλουν οι Εστονοί αλλά δεν διατίθενται οι Λετωνοί. Εν πάση περιπτώσει κάπως πρέπει να αναπτυχθεί αυτή η προσπάθεια και για άλλη μια φορά η θέση της Πολωνίας για το όλο αυτό πλέγμα, θα ήθελα να μάθω ποια είναι, για δε τη διασύνδεση με το Ελσίνκι και μετά από το Ταλίν μέχρι το Ελσίνκι, όχι μέσω της Αγίας Πετροπολής, απευθείας, πώς προχωράει. Ευχαριστώ πολύ, Μάικο. Άλλο ένα σημείο που θέλω και εγώ να διατυπώσω, που σε τελευταία ανάλυση αποτελεί συνέχεια στα όσα είπε ο κύριος Κρέμερ. Ως μεγάλος υπέρμαχος των σιδηροδρομών. Έχω σοβαρές επιφυλάξεις προς την δυνατότητα της Πολωνίας να βελτιώσει την κατάσταση στον τομέα των συνδυοδρομικών μεταφορών. Ερωτώ λοιπόν, όπως και ο Μιχαήλ, είναι διατεθειμένη η Πολωνία να κάνει και το δικό της μερίδιο της δουλειάς στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Και αυτό χωρίς να μπούμε στα πολύ βαθιά πολιτικά νερά βέβαια. Φοβάμαι πρόεδρε ότι αν διστάζαμε να μπούμε σε πολιτικά ύδατα δεν θα, δεν θα έβλεπε ποτέ το, το, το φως της ημέρας η Βία Ξεκινώ πάντως λέγοντας ότι υπάρχουν και θα μπορούσαν να υπάρξουν πολλά ερωτηματικά. Τα είχα και εγώ όταν ξεκίνησα και ανέλαβα τη θέση αυτή. Εάν Δεν τα απαντούσε ωστόσο, νομίζω ότι ούτε τη δική μου, το δικό μου χρόνο, ούτε το χρόνο της κυβέρνησης θα σπαταλούσε εδώ πέρα. Κατάλαβα τώρα που σας άκουγα, προσπάθησα να ακούσω διερμηνία, αλλά τελικά κατάλαβα και τι λέτε χωρίς, να σας, ε, χωρίς διερμηνία. Να ξεκαθαρίσω κάτι για την ε, κατάσταση στην Πολωνία. Όταν ξεκινήσαμε τον James, οι πιο δύσκολες συζητήσεις που είχα ήταν στην Βασοβία. Μας είπαν σαφώς δεν είναι προτεραιότητα για μας. Έχουμε άλλες προτεραιότητες. Ανατολή-Δύση, άλλα έργα, που εντάξει, δικαίωμά του. Αλλά θεωρήσαμε ότι ήταν σημαντικό να καταλάβει και η Πολωνία ότι υπήρχε ένα βαθμό αλληλεγγύη τη της Ευρωπαϊκή Ένωση με την Πολωνία και οικονομικά και θα περιμέναμε και να μην είχε η Πολωνία το βαθμό ενδιαφέροντος για το έργο ε, που είχαν άλλε χώρε να έδειχναν κάποια αλληλεγγύη και αυτές με τη, Βαλτική, με τη Βαλτική. Σήμερα μπορώ να σας πω ότι υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη και μπορώ να σας πω χωρί να είμαι Πολωνό, ότι μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική, αλλά πάντω μέχρι σήμερα δεν θεωρούμε ότι θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα από την Πολωνία. Να πω στον κύριο Σάντα ότι έχουμε επιστολές από την Ανατολική Πολωνία που τονίζουν την σημασία της, ε, του Rail Baltica ακριβώς για τους λόγους που αναφέρατε ότι υπάρχουν, έχει μόνιμο η συμφόρηση των οδικών μεταφορών εκεί και ζητούν συνδρομικές μεταφορές. Αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πραγματική σύνδεση με το τρένο μεταξύ Ταλίν και Βασοβίας. Αν θέλεις να φορτώσει ένα τρένο με εμπορεύματα στο Ελσίνκι, στο Ταλίν. Για να φτάσει στην Πολωνία θα πάρει χρόνια. Μία μέρα ε, ε, είναι, ε, κρατάει αυτό το απειρχιωμένο σύστημα φωτοεκφόρτωσης η Rail Baltica μπορεί να αλλάξει την επιχειρηματική κατάσταση. Η ερωτή σας κύριε Σάρα για μας αυτό που έχει σημασία είναι να συζητούμε με τις επιχειρήσεις και να δούμε την, τις δυνατότητες της Rail Baltica. Η απάντησή μου είναι ότι υπάρχουν δυνατότητες αλλά προφανώς η επένδυση είναι μεγάλη. Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν υπάρχουν τα λεφτά. Θα μπορούσαμε να το δούμε σαν μια ενδιάμεση λύση για τις οδικές μεταφορές. Μπορεί να υπάρχουν επιβατικές μεταφορές σε ένα κομμάτι στην Πολωνία γύρω από τη Ρήγα, αλλά όχι σε όλη τη χώρα. Και μην ξεχνάτε και, τις, και τα μεγέθη, ας πούμε. Όλος ο πληθυσμός της, ε, των βαλτικών χωρών είναι μικρότερος από της Τσεχίας. Αυτό που θεωρούμε είναι ότι η Rail Baltica θα αλλάξει τη δυναμική των μετακινήσεων. Θέλουμε να συνδέσουμε και με την ε, Βίλνα. Θεωρούμε ότι είναι σημαντική επένδυση με την Βάλκα. Βάλκα και θα παίξει ρόλο και στην ε, ανάπτυξη της Λετωνίας. Τώρα, η οικονομική βιωσιμότητα του Ευρωπαϊκού Εύρους Γραμμής. Η μελέτη αποτελεσματικότητας πριν από 3,5 χρόνια έλεγε ότι η επένδυση για ένα τρένο για μια γραμμή ευρωπαϊκού εύρους μέχρι, την, ε, μέχρι το Ταλίν θα κόστισε 3 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι αδύνατο. Κάναμε μια προσέγγιση βαθμιαία, εξετάζοντας προσεκτικά την κατάσταση των γραμμών σήμερα. Σας είπα κάπου στην παρέμβασή μου ότι σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο να μετακινήσουμε την το ρωσικό εύρο γραμμή κατά κάποια εκατοστά και να, τη μία, δηλαδή, τη μία ράγα για να φτάσει στην, ε, στο ευρωπαϊκό. Και ότι αυτό θα έχει μικρότερο κόστο. Θα προχωρήσουμε σταδιακά. Αλλά η απάντηση να κάνουμε την Rail Baltica ευρωπαϊκού εύρος γραμμή τώρα θα σα έλεγα όχι. Στρατηγικά ωστόσο πιστεύω ότι το εύρος γραμμή πρέπει να φτάσει το ταχύτερο δυνατό στο κάουνα. Βεβαίω θέλουμε τις ιδιωτικέ επενδύσεις, αλλά σήμερα για να σας το πω ομά, δεν υπάρχουν και τόσοι πολλοί οι ιδιώτες που ασχολούνται με τις ιδεοδομικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Οι περισσότερες εταιρείε είναι κρατικές, μεγαλώνουν, ενώ οι ιδιώτες που ασχολούνται με το τομέα και κερδίζουν είναι λίγοι. Υπάρχει ωστόσο ενδιαφέρον για την περιοχή και εξετάζουμε το ενδεχόμενο επενδύσεων. Είμαστε όμως έτοιμοι να στηρίξουμε το ιδιωτικό κεφάλαιο συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα, συμπράξεις ιδιωτικού δημοσίου και ευρωπαϊκών πόρων. Η απάντησή μας είναι ναι. Είναι κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε και έχουμε μερικά ενδιαφέροντα θετικά στοιχεία. Το ερώτημα είναι πότε θα ξεκινήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, αλλά αυτό έχει να κάνει με το θέμα του ελεύθερου ανταγωνισμού και το θέμα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε πολλού πολλούς επιχειρηματίες σε μία χώρα ε, και να συμπεριφέρονται σαν μονοβολιακά. Ιωνή. Κυρία Σαββισάρ. Ναι. Η ιδέα μας είναι 120 χιλιόμετρα την ώρα. Το αν θα φτάσουμε αμέσως ή όχι δεν είναι καταστροφικό και πρέπει να δούμε γιατί είναι πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Δεν θα έκανα απλοποίηση αν έλεγα ότι ε, μειώθηκε η εμπιστοσύνη στο Rail Baltic. Εγώ έχω εμπιστοσύνη. Πιστεύω ότι μετά από χρόνια ε, στα ευρωπαϊκά δεν είμαι και τελείως αφελής. Νομίζω ότι έχουν, έχει μέλλον δεν θα αποκτήσουν, δεν θα αποτύχουν. Μπορεί να προερχόμαστε από μια χώρα που προέρχομαι ξέρετε μια χώρα που ε, στο ξεκίνημα δεν ήμασταν και τρομερά ενθουσιασμένοι, ενθουσιώδεις με την Ευρώπη. Τώρα όμως η Εστονία λειτουργεί καλά. Αν προκύψει βέβαια και στην Εστονία μια κατάσταση αντίστοιχη με την Λετωνία θα το ξαναδούμε. Τώρα, τι θα γίνει με τη συγχρηματοδότηση. Αυτό είναι μία από τις δυνατότητες που μπορούμε να εξετάσουμε. Επίσης μπορούμε να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο ότι τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων των χωρών αυτών. Μήπως θα μπορούσαν οι χώρες αυτές να αναζητήσουν ε, χρηματοδότηση ε, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν νομίζω ότι η κατάσταση βέβαια είναι σε τέτοιο βαθμό που να πούμε ότι χάνουμε την, εμπιστοσύνη, την εμπιστοσύνη μας. Αλλά επιπλέον να σας πω ότι αποτυχία δεν συμφέρει ούτε την Ευρώπη ούτε τις χώρες αυτές. Είναι κρίσιμα, κρί, κρίσιμη οικονομική κατάσταση. Δεν υπάρχουν πολλές πύλες προς Ανατολάς που μπορεί να χρησιμοποιήσουν Ευρωπαίοι, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις εδώ. Νομίζω ότι απάντησα σε κάποιες από σας κύριε Κράμελ. Οδική συμφόρηση, ναι. Γι' αυτό δουλεύω και για το Rail Baltica. Αποτελεί τη μόνη πιθανή λύση για το μέλλον. Σε συνεργασία με τα λιμάνια βέβαια, αυτό το πιστεύω. Δεύτερον, η Πολωνία είναι έτοιμη, νομίζω απάντησα. Πιστεύουμε αυτή τη στιγμή ότι Πολωνία εφαρμόζει αυτά που, που, που έχει, για τα οποία έχει δεσμευτεί. Θα πάω στο εγγύς μέλλον στην Πολωνία. Δεν έχω δει τίποτα το αρνητικό προς το παρόν. Μπορεί να μην χοροπηδούν από τη χαρά τους, αλλά κάνουν τη δουλειά τους. Ήρπιν. Για το Ήρπιν για την ε, για το ευρωπαϊκό εύρος γραμμή. Σας είπα ότι το να φτιάξουμε ένα σιδηρόδρομο με ευρωπαϊκό εύρος γραμμή που θα κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια, θα σας έλεγα όχι. Ωραία ιδέα του να έχουμε το όραμα ενός ε, τρένου υψηλής ταχύτητας με, ευρωπαϊκή, με ευρωπαϊκό εύρος, γραμμή γραμμής από το ε, Ταλίν, αλλά να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Ο στόχος μου νομίζω είναι να φτάσει η το ευρωπαϊκό εύρος μέχρι το Κάουνας. Το για όλη τη Rail Baltica δεν είναι ε, ε, τη στιγμή. Το πώ θα πάει τώρα στο κάουνα από το ΕΡΚ ή όχι είναι άλλο ζήτημα που θα το δουν οι Πολωνοί. Έτσι ο πρώτος στόχος θα είναι πρώτα τουλάχιστον να πάμε μέχρι την ε, το Μαρίενστατ μέχρι το Μόσκαβα για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και την, ε, τις επιχειρήσεις. Αυτά για τις προτεραιότητες μας. Δεν θα σας δώσω ε, ημερομηνίε. Αν με ρωτήσετε, δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένες ημερομηνίε, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και πάντως θα πρέπει το, ο κόμβος να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια. Δηλαδή θα είχε κανένα νόημα να κάνουμε ε, το Rail Baltica και να περνάει μερικά χιλιόμετρα, μερικέ εκατοντάδε χιλιόμετρα μακριά από έναν ευρωπαϊκό κόμβο. Θα πρέπει να συνδεθεί κάπω. Καθώ είμαστε εδώ και κοντά στο αεροδρόμιο, νομίζω ότι δίνονται αρκετέ δυνατότητε και δεν ξέρω αν έχω απαντήσει την ερώτηση. Σα ευχαριστώ. Κύριε Τελικά, ευχαριστώ. Για τη σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας. Και εμείς θέλουμε στο μέρο να σας ξαναδούμε. Και εγώ σας συγχαίρω για την εκλογή σας και καλή εργασία στη, καλές εργασίες στο υπόλοιπο της αιτίας σας. Last but certainly not least, um, and been very patient. Και εν τέλει, περιμένουμε πολύ υπομονή. Ο κύριος Βίνα ως προς το σχέδιο ERTMS. Και θα ήθελα ξεκινώντα να πω ότι με μεγάλη χαρά είδα για το ETCS ότι έχετε κάνει μια σημαντική κίνηση. Δεν ξέρω αν το Ηνωμένο Βασίλειο θα ακολουθήσει, αλλά θαύματα πάντα μπορούν να γίνουν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εφόσον έχω επιφορτιστεί με το σύστημα ERTMS που σχετίζεται με την ταχύτητα και θέλω να επιταχύνουμε τις τι εργασίε μα. Θα προσπαθήσω να το παρουσιάσω όσο πιο σύντομα μπορώ. Στην πρώτη μου εντολή είχα δύο στόχου. Πρώτα απ' όλα να υποστηρίξω την Train και την υπηρεσία, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων για να εισάγω και να καθορίσω τι προδιαγραφέ ETCS. Τι ενιαίε προδιαγραφέ που θα αντικατεστούσαν 23 εθνικέ προδιαγραφέ. Και ήταν το θέμα σηματοδότηση ε, που θα ήταν βασικό στοιχείο της διατουργικότητας. Και σε συμφωνία με τους σιδηροδρομικούς εισεγάγαμε έξι προτεραιότητες, δηλαδή έξι διαδρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων. Θέλαμε οι σιδηρόδρομοι να είναι αξιόπιστη εναλλακτική για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. Γιατί η προτεραιότητα δόθηκε στο εμπόρευμα, στα εμπορεύματα. Καταρχάς χρειαζόταν να καλύψουμε ένα κενό διότι όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, η μεταφορά εμπορευμάτων ήταν πολύ μικρή σε όγκο και θα έπρεπε να μπορέσουμε να συνδεθούμε και με άλλου τρόπου μεταφορά εμπορευμάτων. Και κάτι άλλο που βλέπουμε όλο και περισσότερο, ότι το δίκτυο για τι συνδρομικέ μεταφορέ φορτίων θα μπορούσε να συμβάλλει για την επίτευξη των στόχων τη Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική πολιτική και να μειώσουμε τι αλλαγέ του κλίματο. Τι καταλάβαμε πρώτα απ' όλα και τι έγινε. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να καθορίσουμε ε, κοινό στατηγικό πλαίσιο για του σιδηροδρόμους και αυτό το πετύχαμε μέσω δύο υπομνημάτων συνεννόησης, ένα το 2005, όπου εκεί ε, μοιράστηκε ο ρόλος των διαφόρων ενδιαφερομένων και μετά υπόμνημα που υπογράφηκε το 2007, όπου εκεί καθορίστηκαμε καθορίσαμε πώς θα αναπτυχθεί το ERTMS στους έξι αυτούς διαδρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων. Τι καταλάβαμε. Ότι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία των Σιδηροδρόμων είδαμε ότι κατεβλήθησαν προσπάθειες, μεγάλες προσπάθειες τεχνικής φύσεως και τώρα έχουμε ενιαίες προδιαγραφές ETCS. Αυτό είναι κάτι που θεσπίστηκε το 2008 και είναι η εκδοχή 230 δέλτα, ε, διαλειτουργικές προδιαγραφές. Όσον αφορά τους σιδηροδρόμους, ε, θα βελτιώσουμε την κατάσταση στόχος να έχουμε την εκδοχή 3.0.0 που θα επικυρωθεί το τέλος 2012 και θα λειτουργήσει. Δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει διαλειτουργικότητα πριν από αυτό. Είμαστε διαλειτουργικοί με το 300 δέλτα και θα το βελτιώσουμε. Ε, και μέσω λογισμικού. Επιχειρησιακά έχουμε τρεις, έξι διαδρόμους οι διάδρομοι έχουν αναπτυχθεί με διαφορετικό τρόπο. Ε, προς Γενέβη, Στοκόλμη, Νάπολη, μετά είναι Αβέρπ, ε, Λιόν, μετά Βαλένσια, Βουδαπέστη, Δρέσδη, Κωνσταντίνη στη Ρουμανία και μετά Αμβέρσα, Ρότερνταμ προς τα ρωσικά σύνορα μέσω Βερολίνου και Βαρσοβίας. Από πλευράς επιχειρησιακής, όσον αφορά τον κάθε διάδρομο, έχουμε εισάγει κάποιο οργανωτικό πλαίσιο το οποίο είναι σε δύο επίπεδα. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια διαχειριστική επιτροπή η οποία είναι μια επιτροπή υπευθύνων για τις υποδομές που είναι υπεύθυνη για το διάδρομο, για το πρόγραμμα εργασιών που αναπτύσσεται για κάθε ένα τέτοιο διάδρομο και αυτοί διασυνδέονται και με τους φορείς που χρησιμοποιούν το δίκτυο. δεύτερη επιτροπή είναι εκτελεστική όπου εκεί έχουμε προσώπους των Υπουργείων, των κρατών μελών που από τα οποία διαβαίνει ο διάδρομο, Είναι υπεύθυνη για στρατηγική, είναι για, υπεύθυνη για του νόμου που ισχύουν και είναι υπεύθυνη κατά πολύ για τη χρηματοδότηση. Τι πετύχαμε μέχρι τώρα. Η, για του διαδρόμου α, γ και δ έχουμε, έχουν νομική υπόσταση αυτέ οι διαχειριστικέ επιτροπέ. Και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να συντονίσουμε καλύτερα τα προγράμματα και επίσης να εξασφαλίσουμε μια συνέχεια χρονική, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτή είναι χρονοβόρα διαδικασία η υλοποίηση. Τώρα, ε, έχουμε δύο, μετά από δύο-τρία χρόνια, ξέρουμε ότι αυτή η οργανωτική δομή, και το λένε και υπεύθυνοι για τους διαδρόμους, ότι αυτή η οργανωτική δομή, λέγω, σε δύο επίπεδα, είναι παρκής. Τα περίπλοκα πρόγραμμα μπορούν να λειτουργήσουν. Και μπορούμε, πρέπει, χειριστούμε τρεις πτυχές. Πρώτα απ' όλα, να μην υπάρχουν πλέον συμφορήσεις στις υποδομές. Δεύτερον, να εισάγουμε το ERTMS και τρίτον, θέλουμε να διοργανώσουμε τις λειτουργικές πτυχές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κατά μέσο όρο, το μήκος των σειρμών είναι 440 μέτρα στην Ευρώπη. Μπορεί να αυξηθεί το μήκος χωρίς πολύ μεγάλη επένδυση στα 750 μέτρα και αμέσως βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες βελτιώσεις. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι αν πάρουμε τα τρία στοιχεία, τους τρεις παράγοντες, και είναι και στόχος μας σε κάποιους δρόμους μπορούμε μια αύξηση του παρόντος δυναμικού κατά 50%, 5-0. Όσον αφορά την ασφάλεια και την ακρίβεια των δρομολογίων, θα τα βελτιώσουμε όλα αυτά κατά 20-25%. Άρα μιλάμε για σημαντικές αλλαγές. Και κάτι άλλο το οποίο ήθελα να τονίσω, γιατί αυτή είναι η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει όσον αφορά τη λειτουργία των διαδρόμων αυτών, είναι ότι απαιτείται πολύ σημαντική προσπάθεια συντονιστική Χρειάζεται συντονιστική προσπάθεια πλευρά κατών μελών και από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από του διαφόρου εμπλεκομένου του τομέα των σιδηροδρόμων και από όλο τον τομέα και εκείνου που παρέχουν τον εξοπλισμό κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να τα χειριστούμε. Χρειάζεται συντονισμό των δράσεων, ούτω ώστε τελικά να πετύχουμε τα απαραίτητα αποτελέσματα. Για κάτι άλλο το που θέλω να τονίσω σε αυτή τη φάση, να το πω και να το υπογραμμίσω, είναι ότι χρειαζόμαστε μια κοινή ε, εικόνα όσον αφορά το πώ θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Κυρίω από τα κάτι μέλη τα οποία διασχίζει ο διάδρομο, αν υπάρχουν σου καθυστερήσει από πλευρά ενό κράτου μέλου από το οποίο περνάει ε, ο διάδρομο, τότε καθυστερεί όλη η υλοποίηση. Χρειάζεται προσαρμογή, χρειάζεται συντονισμό μεταξύ κρατών μελών, τα οποία συμμετέχουν στο διάδρομο αυτό και τα διασχίζει ο διάδρομος. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν τα μέσα παρακολουθήσεω και εποπτεία για να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα μέσω δύο επιτροπών. Η μία είναι η επιτροπή ERTMS που εξετάζει από τεχνική σκοπιά πώ πηγαίνουν οι προδιαγραφέ και μια επιτροπή, μια ομάδα για το διάδρομο που παρακολουθεί το πώ υλοποιούνται τα συστήματα και πώ εφαρμόζονται στου διαδρόμου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα τον Ιούλιο του ενεστώτος έτου, Στι 22 Ιουλίου εξέδωσε Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Σχέδιο που νημοποιεί αυτού του διαδρόμου μεταφορά εμπορευμάτων και καθορίζει αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή του. Ε, Εξοπλισμό για του σειρμού θα πρέπει να είναι έτοιμο όσον αφορά τη TCS για το 2015 και το 2020 τα αργότερο όσον αφορά του διαδρόμου αυτού και τα διάφορα άλλα υλικά για τις γιατμομηχανές ε, θα λειτουργήσει από 1η Πρώτου 2012 άντε μέχρι 1η Πρώτου 2015. Υπάρχει ένα πλαίσιο. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό για να προωθηθεί το πρόγραμμα. Και ο τομέα το απαιτούσε, ο συνδρομικό τομέα και η βιομηχανία. Θέλαν, δώστε μα, μας λέγανε ένα εργαλείο, ένα μέσο για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε καλύτερε επενδύσει. Τώρα το έχουμε το εργαλείο με το ευρωπαϊκό σχέδιο αναπτύξεως του συστήματος αυτού Ποιε είναι οι προτεραιότητε. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να εφαρμόσουμε την τεχνολογία ETCS, το είπα αυτό, ότι υπάρχουν οι προδιαγραφέ, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι και ο εξοπλισμό που απαιτείται και θα χορηγηθεί από του διάφορου προμηθευτέ ε, θα μπορεί να είναι ε, ανταλλάξιμο, να υπάρχει ισοδυναμία. Γι' αυτό θα υπάρξει ένα σύστημα δοκιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα καθιστά αυτή τη δυνατότητα πραγματικότητα. Μετά το κόστο του νέου εξοπλισμού για το ETCS ε, είναι πάρα πολύ ψηλό θα πρέπει και αυτό να το επεξεργαστούμε για να μειώσουμε την τιμή και το κόστος και έτσι θα δοθεί και κίνητο στους σιδηροδρόμους και πώς θα έχουμε και την έγκριση τελική του 300. Μετά το 2012 θα έχουμε την νόμιμη εκδοχή του συστήματος 3.300. Ποια είναι η βασική πρόκληση όσον αφορά την επόμενη θητεία, αυτή τη θητεία μάλλον. Να μετακινηθούμε από τα εθνικά συστήματα και να πάμε στο ETCS. Και αυτό δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο για τρεις λόγους. Πρώτον, λοιπόν, ε, είναι πολύ μα 30, 40, 50 χρόνια ε, διαρκεί αντέχει ο εξοπλισμός. Και μετά χρειάζεται επένδυση για την αντικατάσταση των σειρμών, των βαγονιών κλπ. Όλα πληρώνται με τριτή σήμερα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και και ειλικρινά να πω ότι κάποιες μεγάλες χώρες διστάζουν δεν λέω ότι δεν θέλουν, διστάζουν όσον αφορά την αλλαγή από τα εθνικά συστήματα προς αυτό, διότι θεωρούν την αποδοτικά, αποτελεσματικά τα εθνικά συστήματα και λένε γιατί να αλλάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ασκήσουμε πιέσει ώστε να γίνει η μετακίνηση από τα εθνικά συστήματα στο ETCS. Πρέπει να πω ότι κάποιες μικρές χώρες αποφάσισαν να αλλάξουν και ήδη το έχουν κάνει. Και τρίτη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε για το μέλλον είναι να είναι λειτουργική αυτή η διάδρομη βάσει του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Σχεδίου. Αυτό απαιτεί κι άλλα μέσα που χρειάζονται. Συμπληρωματικά θα παραθέσω κάποια στοιχεία αργότερα, κυρίω όσον αφορά τα τρία πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Να μειωθεί η συμφόρηση, να εισαχθεί το ETRMS και να εναρμονίσουμε τη λειτουργική προσέγγιση. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν από κοινού ταυτόχρονα, διαφορετικά δεν θα αποκομίσουμε τα πλήρη ωφέλη αυτών των προγραμμάτων. Τώρα οι συστάσεις που έχω ως συντονιστής, έχω συμπεριλάβει, είναι εξή. Όλοι θα πρέπει να καταλαβαίνουν τώρα ότι περνάμε μια κρίσιμη περίοδο. Γιατί? Διότι έχουμε μια εναλλακτική, εναλλακτικό τρόπο ε, μεταφορών με τεχνικές προδιαγραφές που λειτουργεί. Ε, και γι' αυτό έχουμε μια εναλλακτική, εναλλακτικό τρόπο μεταφοράς εμπορευμάτων εν συγκρίση με τι οδικέ μεταφορέ. Άρα ή τώρα ή ποτέ. Πρέπει να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε για πολλά χρόνια. Πρέπει τώρα να τα καταφέρουμε. Να εισαχθεί τώρα η μετακίνηση προ το ETRMS είναι κάτι αξιόπιστο, πιστευτό. Υπάρχουν οι τεχνικέ συνθήκε τώρα, τεχνικέ δυνατότητε και έχει καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Ανεψυχιακό Σχέδιο το χρονοδιάγραμμα. Άρα υπάρχει δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Σχέδιο έχουμε αυτά που μας επιτρέπουν να πετύχουμε το στόχο. Έχουμε τρεις σημαντικές προθεσμίες. Η μία το 2012 για τον εξοπλισμό των τρένων και για την εκδοχή 3 2015 για τα συστήματα των τροχιών και του σειρμούς 2020 θα έχει ολοκληρωθεί όλο το πρόγραμμα για τους διαδρόμους. Μετά, δεύτερο, χρειάζεται υποστήριξη όλων των ενδιαφερομένων χρειάζεται μεγάλη συντονιστική προσπάθεια από τα κράτη-μέλη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον τομέα σιδηροδρόμων, από τη βιομηχανία, ούτω ώστε να συμφωνήσουμε επί των σωστών προτεραιοτήτων και να πετύχουμε του στόχου που έχουν καθοριστεί και συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα υλοποίησεω. Και τρίτον, πρέπει να βρούμε συνεκτικό οικονομικό και νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, οι διάδρομοι ή οι οι έξι διάδρομοι, τους οποίους συζητούμε, δεν έχουν εισαχθεί ακόμα στο πρόγραμμα TENTI, θα πρέπει να ενταχθούν για να υπάρχουν κίνητρα να γίνει η αλλαγή θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση, για τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω, το πρόγραμμα για τις υποδομές απαιτεί βελτιώσεις. Είναι το πιο δαπανηρό πρόγραμμα αυτό για την βελτίωση των υποδομών και χρειάζεται σημαντική προσπάθεια των κρατών μελών με την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό θα πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος TEN-T. Το ERTMS μπορεί να συμβάλλει μόνο στην ανταγωνιστικότητα αν δούμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν για τη βελτιστοποίηση των τριών παραγόντων που προανέφερα. Η ενίσχυση της χρηματοδοτήσεως θα πρέπει να εξεταστεί έγιναν δύο διαγωνισμοί στα πλαίσια των 500 εκατομμυρίων που είχαμε στον προηγούμενο προπολογισμό. Χρησιμοποίησαμε τα χρήματα για να εισάγουμε το ETCS και στι τροχέ και στον εξοπλισμό των τρένων. Λαμβάνοντα υπόψη το χρονοδιάγραμμα το 2012, αυτή την προθεσμία είναι πάρα πολύ σημαντική προθεσμία για το εξοπλισμό των τρένων και για την ανάπτυξη του λογισμικού 3.0.0, θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε και τρίτο διαγωνισμό του 2011. Όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο στόχο το 2012-2020 κατά την άποψή μας, η πρώτη εκτίμησή μας είναι ότι εάν θέλουμε να εξοπλίσουμε τα 25.000 χιλιόμετρα τροχιών και τις ατομηχανές όλες που έχουμε χρειαζόμαστε πάρα πολλά χρήματα που θεωρούμε ότι είναι περίπου 5 δις ευρώ, για να σας δώσω μια ιδέα για την προσπάθεια που χρειάζεται. Έχουμε 3.400 χιλιόμετρα που έχουν καλυφθεί, έχουν εξοπλιστεί, θα έχουμε δεκαπλάσια απόσταση μέχρι το 2020. Πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια, τεράστια προσπάθεια, αλλά είναι και μεγάλη συνεισφορά για τον εξοπλισμό των διαδρόμων. Αυτό το θεωρεί ο σιδηροδρομικό τομέας κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν συμπέρασμα, Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι την τελευταία τετραετία μπορέσαμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα οδηγήσουν σε επιτυχία το στόχο μας για την αγορά αυτή των σιδηροδρόμων, του σιδηροδρομικού τομέα. Μπορέσαμε να καθορίσουμε τις προδιαγραφές, ενίες προδιαγραφές, αντί να έχουμε 23 ξεχωριστές προδιαγραφές που σήμερα ισχύουν. Και δημιουργήσαμε τις κατάλληλες συνθήκες αλλά ήταν μεγάλη πρόκληση αυτή και πρέπει να προχωρήσουμε και να εισαγάγουμε και να εφαρμόσουμε τις προδιαγραφές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για τη συνεργασία τους, τη Γενική Διεύθυνση Τρέν, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Σιδηροδρόμων και τους εκπροσώπους των σιδηροδρόμων. Χωρίς αυτούς θα ήταν αδύνατο να κάνουμε αυτό που θέλαμε, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οι συστάσεις μου είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις για να πετύχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκρός, περάστε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φίνκ. Να μιλήσω γαλλικά. Καλύτερα. Ας μην αρχίσω με προκλητική ερώτηση. Ας μην ρωτήσω δηλαδή αν πραγματικά αξίζει η επένδυση στον κόπο. Νομίζω ότι είμαστε πεπισμένοι όλοι ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα αλλά και με την ασφάλεια. Έχω όμως μια ερώτηση προς τους ρυθμούς της πρόοδου. Θεωρείτε ότι είναι το ζήτημα τόσο τεχνικής, ε, προ, τεχνολογικής προόδου ή υπαρκτών δομών σε παιδοκρατών, αυτό το οποίο καθιστά πιο δυσχερεί την ε, εφαρμογή ή θεωρείτε ότι έχουμε κάποιες δομές επίσης προς την τεχνολογία και τις επενδύσεις. Όταν λέτε ότι υπάρχει κάποια περίοδος ζωής τριακονταετής για την ε, εισαγωγή του συστήματος ε, στους σιδηροδρόμους, μήπως θα πρέπει να συγκεντρωθούμε αποκλειστικά στο refitting, κυρίως όσον αφορά το σαμουά και από εκεί και πέρα ενδεχομένως να διαθέσουμε τα κονδύλια στον τομέα αυτό. Και μια τελευταία ερώτηση. Είτε παλιός βουλευτής είναι κανείς, είτε καινούριο στην Επιτροπή. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κατάλογος προτεραιοτήτων και τα τελευταία χρόνια μάλλον ότι υπάρχει κατάλογος προτεραιοτήτων, ε, βλέπουμε αρκετούς διαφορετικούς καταλόγους προτεραιοτήτων, θα λέγονται δεν αλλάζουν με τον Επίτροπο τόσο όσο με την ε, ε, με τον επαναπροσδιορισμό των στόχων. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να επαναπροσδιορίσουμε τους καταλόγους και τους στόχους όχι συσσωρεύοντας 5-6 διαφορετικούς ε, καταλόγους προτεραιοτήτων, αλλά αν θέλετε να ορίσουμε 5-6-10 προτεραιότητες, μέσα στις οποίες, στις οποίες θα έχουμε και στόχους όμως. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κρέμερ. Αυτή η συζήτηση την έχουμε κάνει εδώ και καιρό και από διάφορες επιχειρήσεις συνδρομικές ακούμε το επιχείρημα πάντοτε ότι είναι ακριβά, χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση, περισσότερα χρήματα, ανεξαρτήτως του πόθεν προέρχονται τα χρήματα αυτά. Εσείς θεωρείτε ότι αρκεί, φτάνει μέχρι εκεί ή μπορούμε να προχωρήσουμε κι άλλο. Και επίσης είχαμε αποφασίσει, το ακούσαμε και σήμερα, ότι υπάρχουν πάνω από 100 διαφορετικέ προτάσει για το πώ θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα συστήματα. Το κύριο όμως χαρακτηριστικό είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει συμβατότητα προ τα άνω και προ τα κάτω, δηλαδή και περαιτέρω να μπορεί να γίνει αναμετατροπή και αναβάθμιση. Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη τη ε, δυνατότητα αναβάθμιση στη συνέχεια, ώστε να μην χρειαστεί όταν έρθει η ώρα να αλλάξουμε και να κάνουμε 25-30 διαφορετικά συστήματα. Επίσης, είναι δεκτόν σε νέες διαδρομές να υπάρχει η εισαγωγή του ΑΕΡΤΕΜΕΣ γιατί θυμάμαι εγώ την περίοδο που φτιάχναμε τον, ε, τροχιά Βερολίνο-Ρόστοκ όπου είχαμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης έχουμε τη χρήση του RTMS σε ένα τούνελ. Υπάρχουν τώρα περισσότερες, ε, περισσότεροι ε, σειρμοί οι οποίοι έχουν εξοπλιστεί με το RTMS προκειμένου να πέρανε μέσα από το τούνελ αυτό του Μπρίνερ. Γιατί βέβαια ξέρουμε ότι πρόκειται για μια στενοπό στην Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν κάποια πρόοδος. Η Ευρώπη έχει μετατρέψει ολόκληρο το σύστημα σε βάση RTMS. Βλέπετε να έχετε τη δυνατότητα να μας εξηγήσετε μια, με μια διεξοδική λίστα, με ένα κατάλογο πού ακριβώς έχει αναπτυχθεί αυτό το σύστημα σε ποιε διαδρομέ Ρώμη, Νάπολη, παραδείγματι είναι στηριγμένοι στο σύστημα του RTMS και σε άλλα αντίστοιχα. Έτσι ώστε να είμαστε θέσει να παρουσιάσουμε και στο κοινό και να δούμε και πώ ε, μπορούμε να διατηρήσουμε την πίεση έτσι ώστε να κλείσουν εν τέλει τα κενά που υπάρχουν γιατί δεν υπάρχει παντού ανεπτυγμένο το σύστημα και υπάρχουν διάφορα κενά. Ευχαριστώ. Κύριε Βίνκ, έχω και εγώ μια ερώτηση. Ή μάλλον δύο. Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο είναι τόσο χλιαρός προς το RTMS, η RTMS. Έστω μπορεί να μην αντιτάσσεται στη χρήση του, στην εισαγωγή του, αλλά πάντως δεν συμπράτηκε πολύ ενεργά. Και επίσης, για να συνεχίσω τόσο είπε ο κ. Κρέμερ, στο ζήτημα της κατασκευής νέων τροχιών στο Βασίλειο γίνεται λόγος για ανάπτυξη μιας νέας υδροτροχιάς από τα βόρεια του και ε, ε, μεγάλης ταχύτητας από τα βόρεια του Λονδίνου μέχρι το Μάντσεστερ θα εισαχθεί εκεί πέρα το ERTMS ή μπορεί να χρειαστεί να έχουμε τα παραδοσιακά συστήματα και ο κύριος Φιντάντσα, αν δεν κάνω λάθος το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν θέλετε σας, σας δανείζω το δικό μας σύστημα της ταξινόμηση έχουμε χαμηλό φάσμα. Όσον αφορά τη εισαγωγή του η e e RTMS, είχαμε βαγόνια παλιά Μπορούσαμε να κάνουμε την ανταλλαγή όταν θέλαμε να το νέο σύστημα και να βάλουμε τη νέα τεχνολογία. Έχουμε προχωρήσει περισσότερο σε συγκρίση με τι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε γιατί είχαν παλιώσει πιο γρήγορα τα συστήματά μα. Κάτι για την ασφάλεια. Η δοκιμάστηκε η χώρα μα πριν από μήνε από τραγικό δυστύχημα στο Βιαρέτζο. Και εκείνο το ατύχημα έφερε στην ημερήσια διάταξη, έδωσε την προσοχή στο θέμα τη ασφάλεια συναρμόνιση των διαφόρων διαδικασιών αδειοδότησης όσον αφορά τις μεταφορές εμπορευμάτων της διεθνής σε διασυνοριακό επίπεδο. Η ανάπτυξη που υποστηρίζουμε εμείς ένθερμα του ERTMS σε όλο το ευρωπαϊκό δίκτυο θα μπορούσε να συνάδει με μια ενίσχυση της δικής μας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ιδροδόμου, μια διαδικασία αναρμονήσεως των αδειοδοτικών διαδικασιών μαζί με μεγαλύτερε, περισσότερε δυνατότητε παρέμβαση από πλευρά υπηρεσία για να αναμονήσουμε τι διάφορε διαδικασίε που καθιστούν ε, πιο ασφαλή ε, τη μεταφορά ε, μέσω των σιδηροδρόμων και να είναι και καλύτερη η ροή όσον αφορά τη μεταφορά και των εμπορευμάτων αλλά και των πολιτών και να λάβουμε υπόψη και εκείνους που κατοικούν κοντά στις δρομικές γραμμές. Όλα αυτά θα πρέπει να ταιριάζουν μεταξύ τους και ελπίζω να τα πετύχουμε όλα αυτά και να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ της εργασίας των εισηγητών και των εργασιών και των προσπαθειών που μπορεί να καταβάλει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνδρομών. Ο κ. Μπάτ έχει το λόγο τελευταίος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Είναι γνωστό ότι τα μεγάλα κράτη θέλουν να διαφυλάξουν, να διατηρήσουν τα συστήματά τους, ενώ τα μικρότερα κυρίως απορρίπτουν μια τέτοια προσέγγιση. Ερωτώ λοιπόν, εσείς έχετε, ή μάλλον διαπιστώνω ότι δεν έχετε ασκήσει πίεση στα κράτη. Πώς θα μπορέσετε να επιτύχετε, πώς θα ασκήσετε πίεση, με ποιον τρόπο. Κύριε δεν έχετε το λόγο. Καταρχάς θα απαντήσω στην ερώτηση του κύριου Γκρόσου με οποίος τις δομές τεχνικές πτυχές δεν είναι το πρόβλημα τώρα. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα συνδυασμό δομών και του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε τη σχέση με τα κράτη-μέλη και, του, και τον διαδρομικό κλάδο. Πολλά είναι τα ζητήματα λοιπόν. Έχουμε ως πρόγραμμα ανάπτυξης και έχουμε και χρηματοδότηση στοχευμένη με αρκετά κονδύλια. Στο πλαίσιο του εθνικού προπολογισμού, λοιπόν, πιστεύουμε ότι θα έχουμε αρκετή υποστήριξη. Επιπλέον, δε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιμένουμε κάποια κονδύλια. Αλλά πάντως πιστεύουμε ότι αρκεί η χρηματοδότηση για του διαδρόμου. Αυτά. για, το, ε, για την εισαγωγή του νέου συστήματος ε, στις νέες, στους νέους σειρμούς ασφαλώς δεν θα υπάρχει δυσκολία να πείσουμε τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την υποχρέωση από το employment plan να το πράξουμε αυτό. Και μάλλον θα πρέπει και να κοιτάξουμε το πρόβλημα να συζητήσουμε με τις αστυνομικέ επιχειρήσεις γιατί καθώς προχωράει ο καιρός έχουμε και ζήτημα υποβάθμισης ε, της, ε, των σειρμών τους, του εξοπλισμού τους. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα για τη χρηματοδότηση αλλά με χρή ενός 50% της ανακαίνησης. Το θέμα είναι στο πλαίσιο του προσεχούς προπολογισμού θα υπάρχει αντίστοιχα αυτή η δυνατότητα. Για δε τις προτεραιότητες φυσικά με εντυπωσιάζουν τα μάλατα όσα είπαν όλοι οι συνάδελφοι εδώ για τις ανάγκες, τα σχέδια, τις ε, τεχνικές πτυχές των μεταφορών. Αυτό που μπορώ εγώ να πω είναι ότι σε σχέση με αυτά που είχαμε πριν από 4 χρόνια το 2005, η σύγκριση είναι συντριπτική. Έχουμε ένα σύστημα, τώρα μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε, μπορούμε να το θέσουμε σε λειτουργία. Για τη τελευταία ανάλυση πρέπει οι ε, μεταφορές φορτίων μέσω σιδηροδρόμου να είναι και ε, ανταγωνιστικές. Αυτή είναι η δουλειά που έχει να κάνει ο συντονιστής. Στις προτεραιότητες επίσης βλέπουμε την ανάγκη να εισαχθούν οι διάδρομοι στα TNT, γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε περισσότερη ευελιξία και για την πρόθεση των ε, επενδύσεων. Για τον κύριο Κρέμερ, οι, πληροφορ... οι διαμαρτυρίες που είχαμε στο παρελθόν τουλάχιστον έχουν μειωθεί σημαντικά. Δεν έχουμε ε, προ προς το 120D, 120D, αν χρειάζεται ένα νέο σύστημα κτλ. Το 230D έχουμε τώρα και ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε στο 2300 έως το 2012. Δύο συστήματα τα οποία είναι συμβατά μεταξύ τους και έτσι μπορούμε να έχουμε ε, σε μια τροχιά είτε το 2 2300 είτε το 30D. Άρα υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης προς τα προς, πρόσω και προς τα πίσω. Και δεν είναι υποχρεωμένη κάποια χώρα κατευθείαν να περάσει το 2 2300D. για, ε, για το ζήτημα της χρηματοδότησης ε, των νέων προμηθειών σε υλικό σιδηροδρομικό. Είδαμε από την ε, Σουηδία τουλάχιστον ότι περίμενε από εμά χρηματοδότηση με βάση το πρόγραμμα που είχαμε προσδιορίσει για τους, για διαδρόμους και νομίζω ότι αν, ήμασταν, ή αν θέλαμε να είμαστε αξιόπιστοι ως προς το πρόγραμμα ή την υλοποίηση του προγράμματος θα έπρεπε θα, θα βλέπαμε ξεκάθαρα την ανταπόκριση της επιπτώσεις στο πρόγραμμα. Και βλέπουμε, όπως άλλωστε και η Επιτροπή διαπιστώνει, ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξάγει όλο και περισσότερο το σύστημα ERTMS, ένα σύστημα ανταγωνιστικό, ένα σύστημα αποδεκτό σε αρκετές χώρες και ταυτόχρονα μπορούμε και να επιδείξουμε την εφαρμογή του όλο και περισσότερο. Έχουμε μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στην Ιταλία. Μπορούμε να μιλήσουμε εξίσου και για την κατάσταση στην Ισπανία. Και πάλι επιμένω ότι σημασία εδώ έχει να συνεχίσουμε, να ακολουθήσουμε το deployment plan για τον διάδρομο καταρχάς. Να λειτουργεί σωστά ο διάδρομος να αποδείξουμε ότι ήταν σωστή η επιλογή και μετά να προχωρήσουμε με την εισαγωγή και εφαρμογή του ERTMS και νομίζω ότι βάσει αυτών μπορούμε να προχωρήσουμε. Πράγμα το οποίο θα επιτρέψει και στο ε, φορτίο μας να, να μετακινείται, να μεταφέρεται κατά τρόπο ανταγωνιστικό. Διαφορετικά αμφιβάλλω αν θα παραμείνει ανταγωνιστική η μεταφορά φορτίων από τους δρόμους. Ο πρόεδρος ρώτησε γιατί είναι τόσο χλιαρή η Βρετανή. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται σε ένα, σε ένα έλλειμμα στο σύστημά μας, ένα ελάττωμα του συστήματος τροποντινά. τους διαδρόμους δεν έχει εισαχθεί ε, οι διάδρομοι δεν έχουν εισαχθεί στον τομέα του φορτίου, της μεταφοράς φορτίου ενώ έχουμε το Eurostar από την άλλη για τις επιβατικές μεταφορές. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια εξέλιξη στον Ηνωμένο Βασίλειο και νομίζω ότι υπάρχει και ευρωπαϊκή υποχρέωση για την εισαγωγή ε, ε, σιδηροτροχιών υψηλής ταχύτητας. Για τον κύριο Φιάνσα θα απαντήσω ότι ναι, έχει δίκιο. Και πρέπει τώρα να εξετάσουμε όλες τις ε, επιπτώσεις αγωγής ενός νέου συστήματος σημαντικού και για τις κρατικές αρχές που καλούνται να το εξετάσουν. Και επιπλέον το θετικό εδώ τώρα είναι ότι υπάρχει το σύστημα. Πριν δεν είχαμε σύστημα για να σταθεροποιήσουμε. Τώρα όμως που το έχουμε Νομίζω ότι, ότι από αυτό εξαρτάται και η αξιοπιστία των ε, διαδρόμων. Και έτσι πρέπει να δούμε τις δυνατότητες για εναρμόνιση όχι μόνο των λειτουργικών οδών αλλά και των οδών ασφαλείας. Ε, και έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε, να αυξήσουμε, μίλησα νωρίτερα για 20-25%. Αυτή είναι η προσδοκία μας ως προς το νέο σύστημα. Ο κύριος Μπάχα... Ρώτησε πώς θα ασκήσουμε πίεση. Να σας πω. Το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα Το θέμα είναι ότι τώρα αυτό που έχουμε είναι ένα ε, νομικό πλαίσιο το οποίο έχουν κάνει δεκτό τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να το τηρήσουν. Επομένω, ε, εναπόκειται στην Επιτροπή να εξετάσει σε ποιο βαθμό οι υποχρεώσει οι οποίε έχουν ε, αναλάβει μέσα από το σχέδιο αυτό τα κράτη-μέλη πληρούνται, τηρούνται. Άρα και εμεί βέβαια κοιτάμε, αλλά πρέπει και η Επιτροπή να εξετάσει σε ποιο βαθμό τα μέτρα αυτά ε, γίνονται σεβαστά. Σας ευχαριστώ κύριε Βίνκ για αυτά που μας είπατε. Και όπως όλοι οι άλλοι, και εγώ λέω προσλέπω σε συνεργασία μαζί σας. Και ελπίζω όλοι να πετύχουμε το όνειρο στο εγγύς μέλλον. Θαύματα χρειάζονται κάποιο χρόνο. Αλλά ας προσπαθήσουμε και να δούμε τι θα πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και να δώσω στη βοηθό σας Φίλιξτο προς Ράγμπι ε, πήρε κάποια χρήματα για να βελτιωθεί ο διάδρομος αυτός μεταφορά εμπορευμάτων. Μπορεί να πείσετε την κυβέρνηση να κάνει τα δέοντα. Ευχαριστώ. Στα διάφορα. Τολμάει κάποιος να έχει κάτι στα διάφορα. Αν δεν τολμά κάποιος να θέσει κάτι στα διάφορα, σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι στον μήνα τον Νοεμβρίο, 9 Νοεμβρίου στις 3 το μεσημέρι. Ευχαριστώ όλους για τη δουλειά τους. Γραμματεία, διερμηνής, πέρα συνεδριάσεως. Καλό βράδυ. <laughs>